Chers collègues, je propose de prendre place. Et... Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με το τυχερό σημείο 13 της ημέρας διάταξης. Αν θέλετε να καθίσετε κιόλας θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο 13 της ημέρας της διάταξης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ηλιανά Γιώτοβα για να εξετάσουμε το σχέδιο νομοδότηση στις συνθήκες εργασία των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τίτλος αφήνει διάφορα υπονοούμενα. Όπως ε, κάνει σαφές ο τίτλος λοιπόν πρέπει να γνωμοδοτήσουμε προς την Επιτροπή Γυναικών. Η κυρία Ιώτοβα θα τα πω στα βουλγάρικα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα εδώ και πολύ καιρό. Το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει γονική άδεια, οικογενειακή άδεια, να αντιμετωπιστούν θέματα διακρίσεων και ιδίως για τις γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές ομάδες μειονοτικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση. Τα προβλήματα αυτά δυστυχώς παραμένουν παρά τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν. Οι γυναίκες σήμερα είναι αυτές οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μας. Οι γυναίκες και οι νέες κοπέλες είναι αυτές οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και γνωρίζουν τι συνέπειε τη. Αλλά συγχρόνως δεν είναι και υπεύθυνε για αυτή την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια αξιολόγηση των συνεπειών τη λιτότητα στην αγορά εργασία και ιδιαίτερα για τι γυναίκε για να δει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Χρειάζεται λοιπόν να δοθούν δυνατότητε για εξέβρεση εργασία, εξασφάλιση τη ισότητα των γυναικών στα θέματα του εργασιακού χώρου, πιο ενεργή πολιτική απασχόληση για τι γυναίκε 9 ε, ε, ναι, γυναίκε από 10 εργαζόνται τώρα στον τομέα των υπηρεσιών. Η επέκταση τη αγορά υπηρεσιών μπορεί να δώσει περισσότερες δυνατότητε στις γυναίκε. Αυτέ είναι θέσει εργασία που τι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καιρό κρίση. Αυτό προτείνουμε λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδότηση. να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό του τομέα των ε, υπηρεσιών, να το αναπτύξουμε περαιτέρω και να δώσουμε τη δυνατότητα στις εργαζόμενες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του τομέα των υπηρεσιών. Το ένα τρίτο της συνολικής απασχόλησης <clears throat> καλύπτεται από τον τομέα των υπηρεσιών και είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον προστοκόμενο στόχο του 75% ποσοστού απασχόλησης μέχρι το 2020 όπως καθορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές του, της Ευρώπης 2020. Επίση πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη εκμετάλλευση στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στι χαμηλότερα αμοιβόμενε εργασίε που καταλαμβάνονται οι θέσει εργασία αυτέ κυρίω από γυναίκε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προσπάθεια να εξασφαλιστούν ελάχιστα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών, όπω είναι τα τακτικά συμβόλαια και διαδικασίε συλλογική ε, διαπραγμάτευση Επίσης οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα τον οικιακό θα πρέπει να <clears throat> έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχε έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες σε όλα αυτά. Οι γυναίκες λοιπόν εργάζονται πολλές φορές στον οικιακό τομέα ή σε δουλειές οι οποίες έχουν καθαρά επαναληπτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να δώσουμε και μεγάλη έμφαση στο θέμα των μεταναστριών γυναικών που είναι πολλές στον τομέα των υπηρεσιών, πολλές από αυτές εργάζονται χωρίς συμβόλαια, με πολύ χαμηλές αποδοχές και χωρίς προστατευμένα κοινωνικά δικαιώματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία και αυτών των εργαζομένων με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ηθαγενείς εργαζόμενες. θα πρέπει να έχουν και αυτέ τη δυνατότητα αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του. Και ένα από τα προβλήματα που έχουμε να κάνουμε και που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο Απασχόληση είναι η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας που προσφέρονται. Δεν μπόρεσα να καλύψω φυσικά όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την απασχόληση των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών λόγω περιορισμών χρόνου, χώρου, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι επί τη βάση αυτού του εγγράφου μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιε λύσει και αναμένω και τι τροπολογίε των συναδέλφων και τι προτάσει που θα περιέχονται σε αυτέ τι τροπολογίε. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Απασχόληση και η Επιτροπή Γυναικών, όπω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα που να περιλαμβάνουν και νομοθετικέ ρυθμίσει, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασία των γυναικών και ώστε να εκμεταλλευτούμε στο ύψιστο στο βαθμό τι δυνατότητε που παρέχει ο τομέα των υπηρεσιών. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν εάν πράγματι έχει πρόθεση να εγκρίνει νομοθεσία για τα θέματα αυτά για να αντιμετωπιστεί η μαύρη εργασία και η εκμετάλλευση, να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών, ώστε να μπορούν να είναι πιο ελκυστικές οι θέσεις που καταλαμβάνουν στον ε, εργασιακό χώρο. Πρόκειται για νομοθεσία που αφορά το τομέα των υπηρεσιών και οριζόντια νομοθεσία, αλλά εδώ θα πρέπει να επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δρόμο της. Είναι ένα αχανές και πάρα πολύ πολύπλοκο θέμα, αλλά Επίση, πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη να εφαρμόζεται η νομοθεσία σωστά και να μην ερμηνεύεται καταχρηστικά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κορ ε, Κόχ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εισαγωγική της παρουσίαση. Γνωρίζω την προβληματική του θέματος αυτού και το γεγονός ότι έχουμε περιορισμούς στον αριθμό των σειρών και σελίδων σε ένα κείμενο, υπάρχουν τα ειδικά προβλήματα τα οποία πράγματι αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και νιώθουν στο πετσί τους. Και ένα από αυτά φυσικά είναι το θέμα της έλλειψης ισορροπίας ανδρών και γυναικών στον τομέα της ε, απασχόλησης. Ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο κείμενο και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι για τα θέματα και τις συμβουλές που θέλουμε να δώσουμε από τη δική μας Επιτροπή. Νομίζω ότι τα κύρια σημεία έχουν όλα αντιμετωπιστεί από την εισηγήτρια και το έγγραφο της Επιτροπής ε, Γυναικών θα έχει δυνατότητα να διεξέλθει αυτά τα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερη έκταση. Νομίζω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας καλύπτει τα ουσιώδη, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ένα σημείο και θα ζητούσα ίσως να υπάρξει περισσότερη συγκεκριμενοποίηση στο κείμενο. Είναι το σημείο 2, όπου αναφέρονται οι φορολογικές ρυθμίσεις και απαλλαγές. Και στο σημείο αυτό εγώ θεωρώ ότι πάντα αυτά τα θέματα φορολογικά είναι υπόθεση των κρατών μελών και υπόκεινται στην επικουρικότητα και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ζητούμε μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση για τα φορολογικά θέματα. Μπορεί σε ορισμένε περιπτώσει να λειτουργούν τα πράγματα καλά, αλλά σε άλλε περιπτώσει μπορεί μια τέτοια ρύθμιση να προσκρούσει σε εθνικέ ρυθμίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο. Η κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ότι μου φαίνεται πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση και φυσικά και η έκθεση στην οποία αναφέρεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένας, μια κατάληψη από τις γυναίκες, μια μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών και το οποίο γεγονός έχει και επιπτώσει στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών που όπως γνωρίζουμε πολλές φορές θίγονται πολύ πιο εύκολα από τα αντίστοιχα δικαιώματα των ανδρών που εργάζονται στον ίδιο αυτό τομέα. Θα καταθέσουμε μια σειρά από τροπολογίες από τη δική μας πλευρά, αλλά θα ήθελα από τώρα <clears throat> να αναφέρω ότι εμείς <clears throat> διαφωνούμε ήδη εξ αρχής με την ε, πρόταση να αυξηθεί η ευκαμψία και η ευελιξία στον εργασιακό χώρο γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ε, η μορφή αυτή της ευελιξίας στον τομέα της εργασίας όταν θίθεται αυτή η ευελιξία ως ο κανόνας και όχι η εξαίρεση η ευελιξία αυτή πάντα αντιμετωπίζεται προς όφελος του εργοδότη και ποτέ σχεδόν του εργαζομένου. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια καλή διάκριση μεταξύ δύο πραγμάτων. Το ένα είναι η ευελιξία της εργασία αιτήσει τη γυναίκα η οποία εργάζεται, διότι θέλει με τον τρόπο αυτό να συμφιλειώσει καλύτερα την εργασιακή τη ζωή με την οικογενειακή τη ζωή. Αλλά είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι η επιβολή από την πλευρά του εργοδότη <clears throat> ευελιξία στην εργασία για του εργαζομένου και συγκεκριμένα για τις γυναίκες, κάτι το οποίο απορριθμίζει απόλυτα την οικογενειακή της ζωή. Είναι δύο διαφορετικά θέματα και αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα συνήθως είναι το δεύτερο, είναι η επιβολή από τον εργοδότη. Επομένως εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχουν σταθερά συμβόλαια με σταθερά ωράρια εργασίας και όντας αυτός ο κανόνας ετήσει της εργαζόμενης γυναίκας για λόγους οικογενειακής ζωής να μπορέσει να ευκαμπτοποιηθεί αυτό το συμβόλαιο. Να μην υπάρξει όμως σύγχυση με την άλλη κατάσταση τη επιβολή από τον εργοδότη, γιατί είναι διαφορετικές καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Η κυρία Ντέλη. τα πρώτα θύματα της κρίσης είναι οι γυναίκες. Σε επαγγέλματα που σε γενικές γραμμές ε, παρουσιάζουν ε, δυσκολίες. Υπάρχει και το θέμα ε, της κακής κατάστασης στην ε, δουλειά, είτε ε, για λόγους ε, σωματικούς είτε για λόγους ηθικούς και πολλές φορές το αποτέλεσμα στην εργασία είναι πάρα πολύ άμεσο. Ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι παράγοντες έκθεσης σε επικίνδυνα σε επικίνδυνες ουσίες, ε, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας. Γιατί γυναίκες που βρίσκονται ε, σε ηλικία αναπαραγωγική δεν πρέπει να ε, έρχονται σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες και επικίνδυνο εξοπλισμό και νομίζω ότι όταν μιλάμε για συνθήκες εργασίας πρέπει να μιλάμε και για την αξία αυτής, δηλαδή πώς ε, εκπληρώνουν, εκπληρώνουν τους στόχους τους ε, οι γυναίκες σήμερα στο χώρο εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει άμεση σχέση με τις συνθήκες εργασίας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να προβλέψουμε τα προβλήματα αυτά με πραγματικές πολιτικές πρόληψεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα κανείς άλλος δεν θέλει να πάρει το λόγο, οπότε ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Γιωτόβα για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους και περιμένω και τις τροπολογίες. Το ερώτημα είναι αρκετά περίπλοκο. Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο, το γνωρίζετε. Εγώ θέτω απλώς το πλαίσιο και πιστεύω ότι όλοι μπορείτε να εμπλουτίσετε την έκθεσή μου ώστε να έχουμε στο τέλος μια πολύ καλή έκθεση σε συνεργασία με την Επιτροπή Γυναικών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Προθεσμία υποβολή σε τροπολογιών 4 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε στις 20 Ιουνίου, γιατί θα τις ψηφίσουμε στις 21 Ιουνίου. Επειδή η Επιτροπή Γυναικών θα εγκρίνει τη δική της έκθεση στις 10 Ιουλίου. Έχουμε ολοκληρώσει με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Καλέ, μη φεύγετε. Κύριε, Φα... Κύριε Φάλμπρ, αντί να διακόψουμε... Euh, λοιπόν, κύριε Φάλμπρ, μήπως να μας παρουσιάσετε την αποστολή στο Τωρίνο Επειδή έχουμε λίγο χρόνο πριν την ψηφοφορία, μήπως μπορείτε να μας ε, πείτε ορισμένα πράγματα για την αποστολή. Γιατί ούτως ή άλλως το απόγευμα δεν θα μπορείτε να είστε εδώ την ώρα που το έχουμε προβλέψει. Λοιπόν, 28. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στο Τωρίνο. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Φάλμπρ που βρέθηκε εκ μέρου μα στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική εκπαίδευση στο Τουρίνο. Έχετε το λόγο κύριε Φάλμπρ. Θα ήθελα καταρχήν την επόμενη φορά να είναι πολυπληθέστερα τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης ε, σε αυτή την ε, επίσκεψη. Θα ήθελα να ήταν περισσότερο στην επίσκεψη γιατί το Τωρίνο είναι πανέμορφο. Και δεύτερον, γιατί ο φορέας τον οποίο επισκεφθήκαμε είναι ένας φορέας πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για την εργασία αυτού του φορέα. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής μέλη της Επιτροπής μας δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτός ο φορέας. 20 εκατομμύρια το χρόνο είναι ο προπολογισμό του, 130 εργαζομένου έχει και εργαζόμενε. Όλοι τους έχουν υψηλά προσόντα. Έχετε ενώπιόν σα το υπόμνημά μα για την ε, επίσκεψη αυτή. Ο φορέας αυτός λειτουργεί σε 31 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και ε, όταν είδαμε αυτά τα οποία παρουσιάσαν είναι σαφές ότι εργάζονται και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος για τον οποίο δραστηριοποιούνται και σε αυτές τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλίσουν την κατάρτιση εργαζομένων από τις χώρες αυτές οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να ξεκινήσουν και να εργάζονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τους δίνουμε τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορέσουν να εργαστούν ως εργαζόμενοι και να μπορέσουν έτσι να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες αυτές στις χώρες τους στη συνέχεια για να ξέρουν πώς γίνονται συλλογικέ διαπραγματεύσεις κτλ. Όπως σας είπα προηγουμένως, η πλειοψηφία των ατόμων με τους οποίους συναντηθήκαμε έχουν υψηλά προσόντα. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες. Το μόνο πράγμα τώρα το οποίο μου φαίνεται ότι ελείπει είναι το να υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιοποίηση των επιτυχιών τους αλλά και των αποτυχιών τους διότι σίγουρα υπάρχουν σημεία τα οποία είναι αρνητικά, δεν λειτουργήσαν καλά και εγώ τους είπα να έρθουν, τους πρότεινα να έρθουν στην Επιτροπή μας και να κάνουν μια σύντομη παρουσίαση για το έργο τους όλο περισσότερο, όσο περισσότερη προπαγάνδα τόσο και καλύτερα. Πιστεύω ότι από τα τέσσερα τους τέσσερις αποκεντρωμένους φορείς που χρηματοδοτούνται στον τομέα αυτό, αυτό είναι ο πιο επιτυχημένος φορέας. Κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ επίσης είναι το γεγονός ότι ο φορέας αυτός δεν αντιδράσει σε επικρίσεις όταν εκτοξεύονται επικρίσεις εναντίον ορισμένων χωρέων, χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ξέρετε ότι υπάρχουν επικρίσεις κατά της Ουκρανίας λόγω της κυρίας Τιμοσέγκο, στο Αζερμπαϊζάν λόγω σύλληψης ορισμένων ατόμων. Εδώ το Κοινοβούλιο ήθιστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικρίνει τις χώρες αυτές. Όλες τις χώρες γενικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όταν παραβιάζονται δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε την πάπια. Εξακολουθεί λοιπόν αυτό ο φορέα να δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία και δεν περιορίζονται από τις ε, αναταραχές οι οποίες ξεκινάνε πάντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο για τα θέματα αυτά. Ελπίζω λοιπόν όπως σας είπα η επόμενη επίσκεψή μας να έχει περισσότερη προσέλευση ένας από τους Ιταλούς συναδελφούς ήθελε να έρθει και ήταν, ε, τελικά ήταν άρρωστος, γι' αυτό καταλήξαμε να είμαστε δύο. Εν τέλει, όταν κατέβαινα από το αεροπλάνο, έπεσα και χτύπησα και μου βάλε πέντε ράματα η, η αρμόδια του φορέα αυτού και αυτό με, μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ, συναδελφέ για την αναφορά. Καλή ιδέα και καλή πρακτική θα έλεγα. Να την υιοθετήσουμε. Δηλαδή, πέρα από την γραπτή αναφορά, να ανταλλάσσουμε και απόψεις στους κόλπους της Επιτροπής. Δεν ε, αρκεί βεβαίω ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμα και τα δύο μαζί. Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Από την πλευρά μου ήμουν επικεφαλή αντιπροσωπεία στο Τωρίνο, όπω ίσω το γνωρίζετε πριν από δύο χρόνια, με δύο άλλα μέλη, τον κύριο Σοντόρ και τον κύριο Ελμέρ. Και είχα αισθανθεί ακριβώ τα ίδια πράγματα με εσάς. Το Ίδρυμα αυτό επιτελεί εξαιρετικό έργο. Χάρη στην ποιότητα της Διευθυντρίας, που για μια γυναίκα αφοσιωμένη στο έργο της, η οποία επαναπροσανατόλισε το έργο του Ιδρύματος σε αρτήση των εξελίξεων στις γειτονικές χώρες και στην Μεσόγειο με πρωτοβουλία άλλωστε του Ιδρύματος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερο συνεπτό έτος, πέρσι, οργανώσαμε κοινή συνεδρίαση των τεσσάρων Ιδρυμάτων επί θέματος που μας επέτρεψε να συγκεράσουμε την εμπειρογνωμοσύνη τους. Πιστεύω επίσης ότι τα τέσσερα Ιδρύματα που εξαρτώνται από την Επιτροπή μας ή που ασχολούνται με θέματα από τον οποίο είμαστε αρμόδιοι, διακρίνονται μεταξύ αντιστοίχων ιδρυμάτων. Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά στον τομέα μας, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τα επιχειρηματά μας, χρειαζόμαστε τεκμηρίωση και αυτό γίνεται με τρόπο υποδηματικό. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να είμαστε όλοι πεπισμένοι για το έργο του Ιδρύματος σε καιρό συζήτησης ε, περί προϋπολογισμών, δημοσιονομικών προοπτικών κλπ. κλπ. Όταν το Συμβουλίο πιστεύει ότι όλα τα κονδύλια που δίνονται σε αυτά τα ιδρύματα περιχούνται από το παράθυρο. Το λέω λοιπόν προς τα μέλη μας. Ε, αν θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι, αν θέλουμε να καινοτομήσουμε, Και δί στον τομέα μας πρέπει να πληρώσουμε. Όσον αφορά τον αριθμό των ε, συμμετοχών στην αποστολή αυτή, το μόνο που ζητώ είναι η Επιτροπή μας να έχει το δικαίωμα να διοργανώσει και μια συνεδρίαση στο Τωρίνο. Βεβαίως, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αυτό δεν είναι δυνατόν. και λόγω του αριθμού των μελών μας, τα μέλη μας τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν είναι περιορισμένα, είναι λόγω των γνωστών οικονομικών περιορισμών. Έτσι λοιπόν έχει κατάσταση. Σας καλώ τώρα. Βάσει αυτού του απολογισμού της επίσκεψης και σε αρτήση και της δικής μας σημερινής διάταξης από εδώ και πέρα να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την ε, πυρογνωμοσύνη του Ιδρύματος σε αρτήση των θεμάτων που συζητούμε. Ο καθένας θα δει πώς θα το κάνει αυτό, αλλά ας δείξουμε περισσότερη ευαισθησία, αξιοποιώντας, όπως είπα, το έργο του Ιδρύματος. Παράδειγμα, χθες συζητούσαμε την πολιτική γειτονία είναι ένα θέμα επί το οποίο θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις με εκπροσώπους του Ιδρύματος. Ευχαριστώ και πάλι για τον απολογισμό όπως ε, προείπα. Χάρηκα που συζήτησαμε το θέμα, έστω και αν στριμώξαμε λίγο την ημερήσια διάταξη, αλλά ε, δώσαμε έτσι την δυνατότητα στα μέλη μας να πάρουν μια ιδέα. Λοιπόν, περνάμε. στο σημείο Περνάμε στο σημείο, συνεχίζει η Πρόεδρος. Μια στιγμή. Στο σημείο 14. Και ξεκινούμε και τις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλοι σας τις κάρτες σας. Ελπίζω να έχετε τον κατάλογο ψηφοφοριών. Στο 14, λοιπόν, ψηφίζουμε. Βελτιστοποίηση του ρόλου της εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Έκθεση από την Επιτροπή Ρέτζι, αρμόδια επί της ουσίας. Η συγγετρία κυρία Χρυσμένοβα από τους Φιλελευθέρους. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τεπολογία 1, σέτερ. Υπέρ, κατά, αποχές, 2, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία D. Από τρεις ομάδες υπέρ. Υπέρ. Το καταλαβαίνω, μάλλον το έλκυνε κατά, αλλά πρώτα είμαστε στο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Μπουλόν. Με προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανεί με την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά. Συμβιβαστική 2 παράγραφο 2. Από τέσσερι ομάδε υπέρ. Τρει ομάδε διορθώνει. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 πάλι σε παράγραφο 2. Κυρία Σρόετρ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφο 3. Συμβιβαστική τροπολογία C από τέσσερι ομάδε Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. παράγραφο 3. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 18. Καταπίπτει. Όλες αυτές οι τροπολογίες μέχρι την 24. Τροπολογία 24. Deutsch. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εντάξει, να επαληθεύσουμε την 25 ηλεκτρονικός. Έχετε δίκιο. Όχι, δεν θέλετε. Καλά, εντάξει τότε. Τροπολογία 26, παράγραφος 4, καταπίπτει. 27, Νταρντέν, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 28, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία ή ε, από δύο ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφα 4 και πάλι, τροπολογία 30 με προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 30 και πάλι με την προφορική τροπολογία. Αν δεν διαφωνεί κανείς, ψηφίζουμε την τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, συμβαστική τροπολογία F εκ μέρους 4 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 36 του κυρίου Πουπάκη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 37, εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 του Ουμάνερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική G της παραγράφου 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 του κυρίου Μπουλό με προφορική τροπολογία δεν υπάρχει διαφωνία, οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 43 καταπίπτει, οπότε πάμε στη 44 της κυρίας Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 6, τροπολογία 45 της κυρίας Χάρκιν με προφορική τροπολογία καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε την 46 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο τώρα της γνωμοδότησης ηλεκτρονικός παρακαλώ. Tout le monde a Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψηφίσαντε 42-39 υπέρ, ε, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία του σημείου 16, Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 του κυρίου Αντάμ Κόζα. Παράγραφος 1 του άρθρου 1, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4, παράγραφος 1, Α, να, να, να επαληθεύσουμε την 26 θέλετε. Καλώς. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 υπέρ. 42 ψηφίσαντες. 23 υπέρ και 18 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 1 συμβιβαστική τροπολογία α. α εκ μέρους 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4 παράγραφος 2 3α ε, νέο τροπολογία 30 ρίκα μάνερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 4 παράγραφος 3. Συμβιβαστική τροπολογία β εκ μέρους 4 ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Άρθρο 4, παράγραφος 3, 32, τροπολογία καταπίπτει. Οπότε πάμε στο άρθρο 5, συμβιβαστική C, εκ μέρους 4 ομάδων υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 1, η 37 έχει αποσυρθεί. Οπότε ψηφίζουμε τώρα την 38 της κυρίας Παπαδοπούλου με προφορική τροπολογία. Δεν διαφωνεί κανείς με την τροπολογία την προφορική, οπότε ψηφίζουμε την 38 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 8, τροπολογία 39 της κυρία Καρή Μαντέλη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 Τόμας Χάντελ ε, την ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 έχει αποσυρθεί, οπότε ψηφίζουμε τώρα στο παράρτημα τη 42 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράρτημα τίτλος 1, συμβαστική D, τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική E, από τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 της κυρίας Ντέλη υπέρ. Κατά αποχές ξανά. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 ρίκα μάνε ριπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 ντέλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 και πάλι ντέλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 ντέλη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 ντέλι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 Τόμας Χέντελ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο σημείο 2 τώρα του παραρτήματος, τροπολογία 56 του κυρίου Πουπάκη. Κατά τμήματα ψηφοφορία, τη ζήτησαν οι σοσιαλιστές το σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε εκτός από το end unrest, υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ της προσθήκης του end unrest. rest, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται λοιπόν. 57 Kinga Guns, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 58, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται 6 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 Thomas Handel με προφορική τροπολογία της κυρίας Παπαδοπούλου. Δεν διαφωνεί κανείς. Α! Οπότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της τροπολογίας 59 υπέρ, της αρχικής τροπολογίας λοιπόν, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 Τόμας Χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 Χέντελ υπέρ κατά δεν είναι σε το αποτέλεσμα 61 και πάλι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός να ψηφίσουμε άλλωστε τόση ώρα δεν έχουμε ψηφίσει ηλεκτρονικά Tout le monde a pu voter, le vote. Ψηφίσατε όλοι υπέρα της ψηφοφορίας. 44 ψηφίσαντες, 19 υπέρ 23, 20 υπέρ 23 κατά, δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται. Συμβιβαστική F από 4 ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 63 υπέρ, κατά, Δεν βλέπω τους φιλελεύθερους. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 του κυρίου Ποπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G εκ μέρους τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 ντέλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 Καταπίπτη. άρα πάμε στην 11. Κόζα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 γκέντς υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικό. Στην 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 44 ψηφίσαντες. 18 υπέρ, 23 κατά, ε, δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται. 76 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται και πάλι. Συμβιβαστική H, από 4 ομάδες, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79, Ρίκα Μάνερ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83, Χέντελ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 έχει αποσυρθεί. 81. Χέντελ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 πουπάκι. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Χέντελ λιπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Φραντζ Ομπερμάγερ. Με προφορική τροπολογία. Για την οποία δεν διαφωνεί κανείς. Άρα ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 17. Ντέλη. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 18. Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 19. Χέντελ. Υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Χάντελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Όμπερμαϊερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Όμπερμαϊερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Όμπερμαϊερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοδότησης. ηλεκτρονικός ψηφίζουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι όλες σε πέραση της ψηφοφορίας. 45 ψήφισαν, 41 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. και προχωρούμε. Στο σημείο 17, ε, Προπολογισμό 2013 εντολή για τον τριγωνικό διάλογο. Ο εισηγητή γνωμοδότηση είναι ο κύριος Φιλίπ Μπουλάν. Παράγραφο 1. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 Κάμπρνοχ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 Γιονς, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 10. Ζούμπερ υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία 11 Γκέντς. με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 11 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. Τροπολογία συμβασμού σε. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, ενεκρίθη. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχω κάποια αμφιβολίε για το κατάλογο ψηφοφορία. Ίσως μπορεί να το διευκρινίσει ο εισηγητή. Γιατί έρχεται τη συμβαστική ΔΕ μετά τι τροπολογίε 17 και 18. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, μετά την παράγραφο 4, συμβαστική τροπολογία D, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ναι, ναι, ξέχασα όμως να ψηφίσουμε την τροπολογία 18 της κυρίας Τζιν Λαμπέρτ. Τη ζητώ ταπεινά συγγνώμη. 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά έχουμε ψηφίσει μόνο το τμήμα Not least of elder workers Και τώρα, μετά την παραγωγή 4, πάμε στην τροπολογία 20. Ζουμπέρ με προφορική τροποποίηση, δεν βλέπω αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση. Χωρίς την προφορική τροποποίηση, υπέρ. Δεν έχει γίνει δεκτή η ψήφιση της προφορικής τροποποίησης. Επειδή υπήρξε αντίρρηση. 20 χωρίς την προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 21. Εκπίπτει. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. χωρίς τη φράση θεωρούν ότι η εθνική συνεισφορά δεν πρέπει να ξεπερνάει το 10%. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Το ψηφίσουμε και αυτό. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 της κυρίας Ζουμπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24. Δαρδέν και άλλων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 Πέρας ψηφοφορίες. 45 ψήφισε, 37 υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή μας, του ευχόμαστε καλές διαπραγματεύσεις. Nous en venons au point 18 euh, vers une reprise génératrice d'emploi, euh, adoption d'une question avec demande Σχέδιο προφορική ερώτηση και έγκριση πρόταση ψηφίσματο. Ακολουθώ την εισηγήτρια. Προτείνω να ψηφίσουμε επί τη προφορική ερώτηση πρώτα. Εισαγωγικό μέρο Εκεί έχουμε τροπολογία από το ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επί του ερωτήματος 1 έχουμε δύο τροπολογίες από το ΕΛΚ κατά τη ψηφοφορία. Σχολή εκτός μικροφώνου. Σας είπα, νομίζω ήταν σαφής, σαφές το αποτέλεσμα της προηγούμενης ψηφοφορίας, αλλά αν θέλετε να επαληθεύσουμε για την τροπολογία 1. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν θέλει το ΕΛΚ, άλλη μόνο. Ψηφίσαμε. Ελπίζω να ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφορίας. 43 ψηφίσαντες, 22 υπέρ, 20 κατά. Είχατε δίκιο. Ήταν πολύ κοντά. Καλά κάναμε και πάλι Εγκρίνεται πάντως. Ερώτηση 1. Τροπολογία 2. ΕΛΚ κατά τμήματα. Τμήμα 1. Ψηφίζουμε. Από το what does μέχρι το setting systems. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τμήμα 2. Αν εγκριθεί θα αποτελέσει επιπλέον ερώτημα. Υπέρ. Κατά αποχές. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται ως επιπλέον ερώτημα. Εν συνεχεία, τροπολογία 3, καταπίπτει. Α, με συγχωρείτε. Όχι, ψηφίζουμε για την 3 ξεχωριστά, υπέρ, κατά, αποχές, αεγκρίνεται. Παράγραφος, μάλλον ερώτημα 4, τροπολογία 4, L από, το, από φιλελευθέρους, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί του συνόλου της, ε, προφορικής ερώτησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαμε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. δεν ψηφίσαν ψηφίσαντων. Τρεις εποχές ένας κατά εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα επί της πρότασης ψηφίσματος. Παράγραφος 1, συμβαστική, β, τριών ομάδων υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα. Α, να επαληθεύσουμε. Επί της συμβαστικής β. Ψηφίζουμε. Ψήφισαμε όλοι. Πέρας ψηφορίας. ψηφορία. 21 υπέρ, 17 κατά δύο εποχές. Εγκρίνεται όντως. Τροπολογία 22 των πρασίνων υπέρ. Κατά εποχές. Εγκρίνεται. 23 σοσιαλιστές υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 πράσινη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 των πρασινων με προφορική τροπολογία αν δεν υπάρχει αντίρρηση ψηφίζουμε υπέρ κατά οι φιλελεύθεροι δεν ψηφίσουν 25 υπέρ και πάλι κατά αποχές να επαληθεύσουμε παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Αν ψηφίσαμε πέρας ψηφορίας. 42, μάλλον 18 υπέρ, 16 κατά, 6 εποχές. Εγκρίνεται. Πράγμα 2. Συμβαστική σε τριών ομάδων υπέρ, κατά, εποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. 30 ε, σοσιαλιστές υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 των φιλελευθέρων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 φιλελεύθεροι με προφορική τροπολογία της ίδρυας, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, υπέρ, είναι 32, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. 33 συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πράγμα 4. 34 από τους πράσινους υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 των σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Ξέχασα την 35 του ΕΛΚΑ. Ζητώ συγγνώμη. Υπέρ. Κατά αποχές. εγκρίνεται. Παραδοσ 5. Συμβαστική δε τριών, μάλλον τεσσάρων ομάδων. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. πράγμα 6. 40. ECR υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41. Ελκ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 του ΕΛΚ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. πράγμα 8, συμβαστική ε, ε, τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 σοσιαλιστών που μπορούμε να προσθέσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε, μετά την παραγραφή 8, έχουμε την 48 της ECR, ψηφίζουμε κατά τμήματα, αποζήτησης ζήτησαν οι Τμήμα πρώτο, χωρίς τις λέξεις του address κλπ. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε. Ψήφισαμε όλοι. Πέραση ψηφορίας. 21 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιο θέλει τώρα να προσταθούν οι λέξει που δεν ψηφίσαμε υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 49 σοσιαλιστών υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. 50 σοσιαλιστών υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. 51 σοσιαλιστών με αίτηση κατά ψηφοφορία από του φιλελευθέρου. Πρώτο τμήμα χωρίς τις λέξεις and to extend μέχρι employment status υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ποιος θέλει να προσθεθούν τώρα οι λέξεις κλπ, κλπ. Ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 σοσιαλιστών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην νέα συμβαστική F δύο ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, 55 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10, 56 ελκ υπέρ κατά αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική για την 56 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσαμε όλοι, Πέραση της ψηφοφορίες. Είκοσι τρεις υπέρ, δεκαέξι κατά. Εγκρίνεται. Και έχουμε και την 59 πέρα των σοσιαλιστών υπέρ. Κατά αποχές Ποιο είναι υπέρ τη 59. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ. 21 κατά. Μία εποχή. Απορρίπτεται. 60 στην παράγραφο 13. Ελκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14, συμβαστική H, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 των πρασίνων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 16, συμβαστική Y, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16, η 66 του ΕΛΚ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17, 67, σοσιαλιστών υπέρ. Κατά, απόχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 19, συμβαστική J, τρεις ομάδε υπέρ. Κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 18, τροπολογία 69, ΕΛΚ υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 19, συμβαστική K, Πέντε ομάδε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα Σοσιαλιστέ με προφορική τροπολογία των ελευθέρων. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε για την 72. Δεν υπάρχει αντίρρηση για, την, για προφορική τροπολογία. Όχι. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη 72. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε την ένα των σοσιαλιστών μετά. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Στο προημείο συμβαστική α τεσσάρων ομάδων τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΠΡΕΜΙΟ Β, 5 ECR υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΠΡΕΜΙΟ D, μάλλον να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα για την 5. Τροπολογία συντηρητικών μεταρρυθμιστών, συντηρητικών μεταρρυθμιστών Εκτό μικροφώνου πρόεδρος. Σχόλια εκτός μικροφώνου και πάλι. Λοιπόν, αποτέλεσμα 18 υπέρ, 23 κατά. Η τροπολογία υπερθυμών 5 απορρίπτεται όπως το είχα ήδη ανακοινώσει. Η έξι τώρα σοσιαλιστών υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Προήμιο F, τροπολογία 9, ΕΛΚ και 8 των φιλελεύθερων. Πρόκειται για ταυτόσημες για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι πέραση τη ψηφοφορία. 43 ψηφίσαντε. 21 υπέρ, 20 κατά. Δεν εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 των σοσιαλιστών υπέρ. Mais monsieur Horry, depuis le début, et comme d'habitude, je n'ai pas ma carte. Κύριο Σωρή, δεν έχει την... Ε, Α, δεν, έχω, δεν έχω την κάρτα της ψηφοφορίας μου το, από την αρχή της ε, ψηφοφορίας και έτσι κάθε φορά που υπάρχει ε, ισοπαλία... Το είπα από την αρχή. Το είπα από την αρχή. Κάθε φορά προσθέτω μία ψήφο κάπου, δεν το έχετε προσέξει. Πού euh, Τροπολογία 10 από την ομάδα των σοσιαλιστών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 από την ECR. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα παραμένει το εκτιμώντας ε, του F. Μετά πάμε στη 12 των φιλελευθέρων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 σοσιαλιστές υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 16 τη CCR. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 του ΕΛΚ. Με προφορική τροπολογία. Της εισηγήτριας. Δεν διαφωνεί κανείς. Άρα ψηφίζουμε τη 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 του ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 του της ΙΑΡ υπέρ κατά υπέρ πάλι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά. Τη 19. Την τροπολογία 19. Του μόνο να Πέρα τη ψηφοφορία. 43 ψηφίσαντες. 22 υπέρ. 15 κατά. 4 αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του σχεδίου ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43 ψηφίσαντες, 36 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στους συντονιστές που συμμετείχαν σε αυτό το ψήφισμα. Πάμε τώρα στο σημείο 19. Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία Έκθεση της Ρίκας Μάνερ. Είναι μια γραμμοδότηση προς την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Η σοσιαλιστική ομάδα θα υπερψηφίσει όλες τις τροπολογίες. Αν έχει, δεν, έχει, δεν έχετε λοιπόν μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί ομού. Όχι, όχι. Ναι, αλλά θα πρέπει να πεις και τους άλλους σοσιαλιστική ομάδα, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά από χες 16 υπέρ κατά απόχες να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι Πέρας. Σαν τα δύο ψήφισαν, 23 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Και δύο αποχές βέβαια. Το πολύ 17 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 εκπίπτει 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω 22 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας δύο ψήφισαν, 20 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 23 των πρασίνων υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 2, <clears throat> υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 3, υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 πάντα σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 8 με προφορική τροποποίηση. Δεν βλέπω αντίρρηση. Ψηφίζουμε την 8 όπως ε, έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά <clears throat> εποχές δεκτή. 9 εκπίπτει. 10 και τελευταία των σοσιαλιστών ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και εδώ δεν έχουμε τελική ψηφοφορία, ήταν απλώς οι τροπολογίες. Και τέλος πρέπει να ψηφίσουμε στο σημείο 15 λέει η πρόεδρο τη γνωμοδότηση της κυρίας Σιλβάνας Ράπτη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας. Συμβαστική τροπολογία F από τρεις ομάδες. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική τροπολογία G τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική E υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 Steinbrook υπέρ κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 της εισηγήτρες Σύρια Στάινρου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 της εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ναι, ναι, θα κάνουμε έλεγχο για την 41. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 17 κατά, γίνεται δεκτή η τροπολογία αυτή. Η 43 είναι συμβατή, ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει 42, περνάμε στην τροπολογία 44. Μια στιγμή λέει η Πρόεδρος. Le 44 est tombé, mais... Η 44 έχει εκπέσει, 45, αλλά και αυτή έχει πέσει. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 13 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Η τροπολογία 48 συμβατή, την ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J, θέτω σε ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 55 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 συζήτητες υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία συμβασμού α ψηφί υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ναι, ναι, μα δεν μπορεί να έχει κανείς ε, μια συμβαστική τροπολογία που να προέρχεται από μια ομάδα και μόνο. Μπας περιπτώσει έχουμε ψηφίσει. 18 καμπνόχ ψήφιπερ. Κατά απόχες απορρίπτεται. Έλεγχος για 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 39 ψήφισε, 18 υπέρ, 19 κατά, δεν γίνεται δεκτή. 19 πιζότο υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική τροπολογία. είναι η τροπολογία 20 με μια προφορική τροπολογία. Δεν είναι συμβαστική τροπολογία, λέει η πρόεδρος. Συμφωνείτε. Είναι η τροπολογία 20 με μια προφορική τροποποίηση, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσουμε, εν πάση περιπτώσει, συμβαστική τροπολογία Β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 πουπάκι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 στάιροκ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 ΚΑΜΠΝΟΧ υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 που πάει υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική τροπολογία σε <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή Θέλετε έλεγχο. Άντε, ας ελέγξουμε. Συμβαστική τροπολογία σε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Γίνεται δεκτή πράγματι. 19-15. Ψηφίζουμε. Συμβιβαστική. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία συμβιβασμού. Φασική τροπολογία D. Υπέρ αποχές δεκτή. 31. Κορνέλσεν υπέρ κατά αποχές Έξι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 32 τροποποιημένη η οποία αναφέρεται στη συμβαστική τροπολογία ε. Αποχές δεκτή. Το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Έχουν κλείσει ψηφοφορίες και σας ευχαριστώ.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 Παρακαλούμε αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε να συνεχίσουμε. Με το σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης, να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτριά μας, τη Γιούτα Στάινρουκ, για την παρουσίαση των τροπολογιών επί της ε, έκθεσής της για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινοτομία. Έχετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια. Μερσή, κυρία Πρόεδρε. Μόνο 290 τροπολογίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να <clears throat> ευχαριστήσω τους και εισηγητές για την εργασία, τη συνεργασία μαζί τους και νομίζω ότι όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Πολλές από αυτές τις τροπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε πολλές κοινέ συμβιβαστικές τροπολογίες. Για τις τροπολογίες τώρα, <clears throat> συγκεκριμένα. Ο τίτλος του κανονισμού έχει απορριφθεί από τις πολιτικές ομάδες αλλά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση για το θέμα αυτό. Άλλα θέματα είναι η κατανομή των πρακτικών, των ε, ποσοστών για, ανάμεσα στις διάφορες δράσεις και η προτεραιότητα, η, το αποθεματικό 5% για τις πολιτικές προτεραιότητες. Εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε, αν μιλάμε απλώς για κοινωνικές ε, επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα. Ίσως ε, η συνάδελφος που έχει καταθέσει αυτή την τροπολογία μπορεί σε κάποια άλλη φάση διμερώς να μου εξηγήσει γιατί δεν είναι παρούσα εδώ. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να καλυφθεί αυτό από μια τροπολογία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και είχαμε ήδη μια συζήτηση για το θέμα αυτό. δεν υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες να αφορούν το θέμα της εταιρική σχέσης που είχαμε ήδη συζητήσει με τους εισηγητές, με τους σκιώδες εισηγητές και ελπίζω ότι και εκεί θα υπάρξει υποστήριξη όλων των συναδέλφων. Ακόμα θέλω να πω κάτι για, τις, ε, για τα τρία ή τέσσερα υποπρογράμματα, καταρχήν για το Progress. Υπήρξαν καλές προτάσεις για μέτρα τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν περαιτέρω από το Progress. Η πρόληψη στον τομέα της ασφάλειας της εργασίας, η συνεργασία μεταξύ σχολείων και κέντρων περαιτέρω κατάρτισης για το όηρες γιούρες. Πιστεύω ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων να ζητήσουμε να υπάρξει πιο ποιοτική εργασία. Υπάρχει το πρόβλημα του brain drain, της απώλειας εγκεφάλων, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί με τα προγράμματα κινητικότητος. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η κινητικότητα δεν πρέπει να οδηγήσει στο να υπάρξει μια μακροχρόνια απομάκρυνση των καλύτερων μυαλών από μια χώρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την υποστήριξη που μου έχουν δώσει οι σκιώδεις εισηγητές για εταιρικές σχέσεις ένθεν και εκείθεν των συνόρων. Πιστεύουμε ότι οι εταιρικές σχέσεις αυτού του είδους θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλύτερη κινητικότητα της εργασίας με συμφωνία των εμπλεκομένων φορέων και επιχειρήσεων και θα πρέπει επομένω να υποστηριχθούν από το πρόγραμμά μας γιατί το κοινωνικό ταμείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει τέτοιου είδους ε, συνεργασίες Έχω ζητήσει λοιπόν από διάφορους συναδέλφους και στις χώρες τους να επισημάνουν αυτό το πρόβλημα. Και πράγματι και αυτοί μου είπαν ότι σε πολλά κρατη κράτη-μέλη υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει αναφερθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη αυτών των εταιρικών σχέσεων σε διαμεθοριακό επίπεδο να υποστηριχθούν από το Κοινωνικό Ταμείο. Μικροχρηματοδότηση και κοινωνικές επιχειρήσεις τώρα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που βασίζονται στην έννοια της κοινωνικού χαρακτήρα επιχείρησης. Αυτό όμως θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο λεπτομεριακά και με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχουν διαφορές απόψεων σε σχέση με την έκθεση παρακολούθησης της Κομισιόν, αν θα είναι ετήσια ή θα γίνεται κάθε δύο χρόνια. Και εδώ μαζί με, με την Πρόεδρο <clears throat> και τους σκιώδης εισηγητές προσθέσαμε ένα τέταρτο άξονα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρξε μια ευρύτατη υποστήριξη στο θέμα αυτό και έγινε σαφές αυτό και από την Ολομέλεια. Αυτός ο άξονας θα πρέπει να μην αφαιρέσει πόρους από τους προηγούμενους τρεις άξονες που έχουν γίνει δεκτοί, αλλά αντίθετα έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί αυτό στο τέταρτος άξονας αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε χωριστή χρηματοδότηση και φυσικά εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας των νέων. Έχω προτείνει τώρα στο τέλος και ένα νέο οριζόντιο κεφάλαιο στον κανονισμό που πρόκειται για τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της Κομισιόν και τη δημιουργία ενός στρατηγικού φορέα ε, διαβούλευσης για τα θέματα αυτά, το ΕΣΥ πρέπει να έχει ως νέο πρόγραμμα και μία προσθέμενη αξία. Πρέπει τα προγράμματα αυτά λοιπόν να έχουν χωριστό, χωριστή δομή λήψης απόφασης και να μην βρίσκεται στην ίδια αιγίδα με τα άλλα προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη λειτουργία του προγράμματος αυτού. Προτείνω επίσης μια σειρά από μέτρα για την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν για τα προγράμματα αυτά και αυτό είναι μια κοινή διεκδίκηση και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου μάλλον για τα θέματα αυτά Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν κινείται προς την, κατή, προς την σωστή κατεύθυνση και δεύτερο έχω ζητήσει να υπάρξει όπως είπαμε αυτός ο στρατηγικός φορέας διαβούλευσης και εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι στην σύλληψη, στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Υπάρχουν τέτοιου είδους δομές στο κοινωνικό ταμείο ή σε άλλα διαφθορτικά ταμεία μετά από τις πρώτες διαβουλεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σε σχέση με τη δομή των προγραμμάτων και η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε εύρωστες συμβιβαστικές λύσεις για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ακόμα ένα ανοιχτό θέμα βέβαια, εκρεμές θέμα με την Κομισιόν. Ίσως θα μπορέσει να μου απαντήσει αργότερα η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ και Σουέτερ. Ευχαριστώ Γιούτα. Έχουμε εργαστεί ήδη και στο παρελθόν για τα θέματα αυτά και για τις τροπολογίες υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπου χρειαζόμαστε ακόμα περαιτέρω επεξεργασία για να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις. Εγώ βλέπω κάπως και τα γρανάζια αυτών των θεμάτων, αλλά κυρίως με νοιάζει το κατά πόσο αυτά θα λειτουργήσουν προς όφελος των ε, τελικών αποδεκτών. Πολλές από τις τροπολογίες μου λοιπόν έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι θα πάει πράγματι το χρήμα στους δικαιούχους και θα γίνει μια διαδικασία η οποία θα έχει απλουστευτεί. Πιστεύω ότι το θέμα των ορισμών είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προσεκτικά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη του να είμαστε προσεκτικοί με τους ορισμούς που θα χρησιμοποιήσουμε. Όταν έχουμε ένα καινοτόμο εργαλείο, δεν πρέπει να μειώσουμε τις δυνατότητες αυτού του καινοτόμου εργαλείου με πολύ περιοριστικούς ορισμούς. πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε να κάνουμε ορισμούς οι οποίοι θα επιβαρύνουν και θα δημιουργήσουν προβλήματα ερμηνείας. Ο κάθε κράτος μέλος, το κάθε κράτος μέλος λοιπόν έχει πολλές φορές διαφορετικό ορισμό, γι' αυτό είναι ένα δύσκολο εργαλείο και επομένως εφόσον είναι καινοτόμο το εργαλείο το οποίο θέλουμε να προωθήσουμε θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτητα στους ορισμούς αυτούς. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι μια μορφή έκκλησης προς την Κομισιόν. Ακριβώς επειδή είναι κάτι το καινοτόμο αυτό το εργαλείο, κάτι το οποίο το επικρατούμε, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να σημαίνει ότι τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής και έχουν καινοτόμο χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ε, χρησιμοποιηθούν με ένα πιο συμμετοχικό τρόπο στο μέλλον. Τρίτο στοιχείο. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει ουσιαστικά μικρές χρηματοδοτήσεις και αυτό δεν πρέπει επομένως να το υπερφορτώσουμε. Ο στόχος μου είναι λοιπόν η καινοτομία η οποία θα προκύψει από αυτό το εργαλείο να μπορέσει να έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και επομένως θα πρέπει να συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικών Θεμάτων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν στενοποί, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα όσμωσης με άλλα εργαλεία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και τον κίνδυνο της διπλής χρηματοδότησης και να να μην κινδυνεύσουμε να χάσουμε προγράμματα τα οποία είναι σημαντικά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα ανοιχτό πλαίσιο και να μην υπάρξουν στεγανοποιήσεις από, από λόγους οι οποίοι είναι καθαρά διοικητικοί. Πρέπει λοιπόν η μικροχρηματοδότηση να μπορέσει να εξασφαλιστεί γιατί αυτό ανοίγει νέες ευκαιρίες και αυτή είναι και η έκκλησή μου προς τους συναδέλφους. Η κυρία Μωρόνς ε, δυστυχώς δεν είναι παρούσα σήμερα, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή προσαρμογή για να καλύψουμε τις ανάγκες των δικαιούχων. Και αυτό αφορά ιδίως το τρίτο τμήμα του προγράμματος που είναι η μικροχρηματοδότηση. Είναι <clears throat> απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο λοιπόν <coughs> θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία της μακροχρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν έχει ληφθεί αυτό στα σοβαρά πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν οι ενέργειες του Κοινωνικού Ταμείου στην, στο να λάβουμε υπόψη την δυνατότητα μικροχρηματοδότησης. Δεν σημαίνει όλα αυτά ότι εγώ βλέπω μόνο τα προβλήματα με τη μικροχρηματοδότηση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε ότι με τόσο μικρές χρηματοδοτήσεις δεν μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε δημόσια στοιχεία, δημόσιο χρήμα προς την κατεύθυνση αυτή αλλά βρίσκεται ακόμα σε ένα επίπεδο δοκιμασίας αυτό το εργαλείο της μικροχρηματοδότησης, οπότε θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να ενισχύσουμε γενικά την προσπάθεια των προγραμμάτων. Κάνω και πάλι μία έκκληση και μία επιχειρηματολογία ώστε να ενισχύσουμε τις εταιρικές σχέσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και δίνει μια ευρωπαϊκή τη θέμενη αξία. Και αυτό δεν αναπόκειται μονάχα στις ε, ευρωπαϊκές αρχές, είναι και θέμα των εθνικών διοικήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει σήμερα για τις διαμεθοριακές συνεργασίες να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια του EURES. και να μην πέσει θύμα στις προσπάθειες ορισμένων εθνικών αρχών να περιορίσουν την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν, στην πράξη να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή χρηματοδότηση για τις εταιρικέ σχέσεις του EURES και να μην θέσουμε εμπόδια και προσκόμματα στη λειτουργία αυτών των εταιρικών σχέσεων, μια τάση που παρουσιάσει και στο παρελθόν και γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω την Κομισιόν να ξεπεράσει τις αντιδράσεις αυτές γιατί ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την πλήρη κινητικότητα των εργαζομένων και στα θέματα αυτά. Κύριε Ντελή, καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνική, η κυρία Σρέτερ τα είπε όλα. Απλώς επί δύο θεμάτων. Δύο πράγματα. Πρώτον, συγχαρητήρια για την εξαιρετική εργασία σε συνεργασία με την κυρία Καταλήξαμε σε συμβαστικές λύσεις. Ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα, δίνει την κατεύθυνση. Πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Ο τέταρτο επίση άξονα πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά το θέμα δηλαδή των νέων. Να καταδικάσουμε την ενεργεία των νέων και χάρη επίση που αναφέρουμε και τον αγώνα κατά της φτώχειας που κατέχει το σημαντικό, το σημαντική θέση εδώ και βεβαίω προσοχή στους ορισμούς, γιατί έχουμε την, την οδηγία για τις υπηρεσίες, έχουμε βέβαια και την ε, κοινωνική οικονομία που αυτή θα μας προστατεύσει σε καιρό Και σπά και μετά ο κύριος Τόμας Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την παρουσίασή της και να τη συγχαρώ για την συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Μόνο σε ένα σημείο θέλω να σταθώ για τα διαμεθοριακά προγράμματα του EURES. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία έχουν ειδικό χαρακτήρα πολλές φορές και πρέπει να εξασφαλιστεί και η συνέχειά τους και να εξασφαλιστεί και η υποστήριξή τους από το Κοινωνικό Ταμείο. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτά τα διεθνικά και διαμεθοριακά προγράμματα για την καιροτομία θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όπως έχει τονίσει και η εισηγήτρια. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία 344, η οποία είναι εύστοχη προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Τόμας Μάν και Μπουλάν το. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Γιούτα. Βλέπεις ότι δεν έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες, δύο-τρεις μονάχα, γιατί ήταν θαυμάσιο το γενικό πλαίσιο. Και υποστηρίζω αυτά που είπε Σρέντερ Πιστεύω ότι το Eures είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να επιληθούν από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της επικουρικότητας. Το κοινωνικό ταμείο έχει πάντα την ανάγκη να σεβαστεί και την επικουρικότητα, αλλά το Eures έχει αυτή την διαμεθοριακή διάσταση που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε μια ουσιαστική και απτή Ευρώπη. Θέλω να κάνω σαφές και στους συναδέλφους ότι στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε μεγαλύτερη κινητικότητα, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να πάνε σε άλλες χώρες εκτός από τη δική τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω θα έχουμε επιδοτήσεις οι οποίες θα μπορούν να κινούνται από 300 μέχρι 1200 ε, ευρώ αλλά φυσικά θα πρέπει να είναι μια επιδότηση η οποία θα γίνεται με επιλεκτικό τρόπο. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη όπου να λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία, εγώ συμφωνώ με την Ελίζαμπε θα πρέπει να είναι δυνατόν να δώσουμε και μια επιδότηση και μια βοήθεια και να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δυνατότητες για τους εργαζομένους να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν πρέπει η Ευρώπη να είναι απλώς ένα κενό γράμμα. Θα πρέπει να έχει σάρκα και οστά. Γι' αυτό συμφωνώ πάρα πολύ με την Ελίζαμπεθ. Δεν πρέπει να πνιγούμε στους υπερβολικούς ορισμούς, θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό πνεύμα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την, το ανοιχτό πνεύμα και την διαφάνεια και εξάλλου δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ταμείο το οποίο έχει άπειρους πόρους, αλλά το ουσιαστικό είναι να εξασφαλίσουμε σωστή εργασία σε επίπεδο περιεχομένου και να επιτύχουμε με τον τρόπο αυτό αυτό το πρόγραμμα παρά το μικρό του μέγεθος να επιτύχει. Και ελπίζω ότι και η Κομισιόν θα, καταναλα... θα καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει και ένας χώρος πειραματισμού αλλά το κυριότερο είναι να μπορέσουμε να έχουμε θετικά παραδείγματα ιστορίες επιτυχίες οι οποίες μπορούν να τύχουν μίμησης. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε αυτό το μικρό πρόγραμμα και να δώσουμε πλήρη έγκριση σε αυτή την έκθεση. Έχει πάρει πάρα πολλές τροπολογίες η έκθεση της κυρίας Στάινοξ, σχεδόν 300, αλλά και αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και επομένω η Κομισιόν θα πρέπει να αποδεχθεί την υποστήριξη αυτού του προγράμματο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν περισσότερη Ευρώπη και μια αυτή η έκθεση κινείται προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πουλά. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ευχαριστώ την κυρία Στάινρουκ για την εξαιρετική εργασία της και για την εξαιρετική συνεργασία με τους Κιώδης και τη συνεργασία εν γέννη. Καταθέσαμε πολλές τροπολογίες συμφωνήσαμε σε πολλές. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σε απασχολήσω περισσότερο. Ε, ίσως το θέμα της ε, και της πρωτοβουλίας για τους νέους ε, εκεί να πρέπει να συζητήσουμε, να συζητήσουμε το ποσοστό κατανομής ενδεχομένως μεταξύ των διαφορών προγραμμάτων και να τονίσουμε το progress και την μικροχρηματοδότηση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι αυτές που δημιουργούν και τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι δεν είμαι κατά της κινητικότητας, το είπε η αλλά δεν ξέρω αν η κινητικότητα είναι αυτή που θα μας λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Στο πλαίσιο του Γιούρες θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τις προσπάθειες εξέβρεσης πρώτης ε, εργασίας και τις διασυνοριακές ανταλλαγές. Όσον αφορά στην Στρατηγική Επιτροπή, μπορεί, ξέρετε, να χρειαζόμαστε την άποψη, τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων στην Επιτροπή αυτή, την Επιτροπή Στρατηγικών Θεμάτων. Δεν ξέρω αν όμως πρέπει όλοι αυτοί να συμπεριληφθούν εκ των προτέρων. Ο Τόμας Μαν μίλησε για καινοτομία πριν από λίγο. Επ' αυτού καταθέσαμε ένα πιλωτικό σχέδιο το οποίο φιλοδοξεί να είναι καινοτομικό με περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινωνική συνοχή. Κάτι το οποίο μας φαίνεται απολύτως απαραίτητο για να τονωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να ενοποιηθεί ακόμη περισσότερο η εσωτερική αγορά. Εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομος και να τονίσω το εξή σημείο. Έχει γίνει σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κίνηση προς την κατεύθυνση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στις ε, απόψεις που έχουν διατυπωθεί προηγουμένως. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω ιδιαίτερα αυτά τα οποία είπε η κυρία Σόντερ και ο κύριος Τόμας Μάνι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση πειραματισμού που ατενίζουμε να δώσουμε ευκαιρίες για καινοτόμες ενέργειες και δεν μπορούμε φυσικά να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία γίνονται. Και πιστεύω ότι θα πρέπει παράλληλα με την εξέταση αυτής της έκθεσης να σκεφτούμε και το γενικότερο θέμα των κοινωνικών επιχειρήσεων και τις δυνατότητες που ανοίγονται για δημιουργικές ενέργειες. Δεν πρέπει λοιπόν οι ορισμοί μέσα στο πρώτο αυτό το άμεσο χρονικό ορίζοντα να είναι ιδιαίτερα περιοριστικοί. Θα πρέπει να δούμε στην πράξη με την πείρα πώς θα είναι ο καλύτερος τρόπος να διατυπώσουμε αυτούς τους ορισμούς και ευχαριστώ και πάλι την εισηγητρία. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Σκόπευα να υποβάλω τροπολογία. Δεν το έκανα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως η συγγήτρια να λάβει υπόψη σε αυτό που ήθελα όταν ε, καταλήξετε στον τίτλο. Διότι μιλούμε για κοινωνική καινοτομία εδώ. Άρα δεν θέλω να δώσουμε την εντύπωση ότι μόνο εδώ συζητούμε το θέμα της κοινωνικής καινοτομίας. Το θέμα αποτελεί ούτως ή άλλως αναπόσπαστο μέρος διαφόρων προγραμμάτων που θα χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό το οποίο καθιστά ιδιαίτερο αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι υποστηρίζει τις κοινωνικές καινοτομίες ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όχι σε κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Οπότε αυτό ακριβώ θα ήθελα να προσθέσουμε στον τίτλο. Δηλαδή την ευρωπαϊκή διάσταση τη κοινωνική καινοτομία. Καταλάβατε. Θα τα ξαναπούμε. Εν πάση περιπτώσει, να μην δώσουμε την εντύπωση ότι μόνο εδώ υπάρχει κοινωνική καινοτομία. Είναι μια διάσταση που, όπως είπα, χαρακτηρίζει και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ, ε, κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν και αν θέλει να λάβει το λόγο. Ναι. Πολύ ωραία, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους τους βουλευτές. Η Κομισιόν στη φάση αυτή έχει λάβει γνώση βεβαίως των τροπολογιών βάσει της αναλυσής της. Πέντε σημεία έχουμε καταγράψει. Το πρώτο διάφορες τροπολογίες διευκρινίζουν το κείμενο ε, υπογραμμίζοντας την κοινωνική διάσταση. Εμείς πιστεύουμε ότι τονίζονταν αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει σημειώνουμε αυτές τις τροπολογίες. Επίσης άλλες ε, νέες προτάσεις έχουν κατατεθεί, νέες ως προς την πρόταση της Κομισιόν. Ακούσαμε και τον τέταρτο άξονα για τους νέους, που δεδομένες τη κατάσταση θα ήταν αφύσικο να απορρίψουμε εννοείται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιπτώσεις. Υπάρχει κάποια επιφύλαξη. Αυτός ο τέταρτο άξονα θα μπορούσε να είναι φυσικά πολύ χρήσιμο, αλλά απαιτεί δυστυχώ και αυτό κάποιο προπολογισμό. Και συναφώς να πω και το εξή. το πρόγραμμα το έχουμε σχεδιάσει στο πλαίσιο του Progress. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε ένα τέρτο άξονα, τι θα γίνει με τους άλλους. Έχουμε και άλλες νέες προτάσεις, νέες προσθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και δει κάτι το οποίο άκουσα σήμερα το πρωί οι διασυνοριακές εργασίε, στα πλαίσια του Γιούρες. Αυτό η Κομισιόν είχε προτείνει να το αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από τη στιγμή πάντως που ένα τέτοιο εργαλείο, ένα τέτοιο μηχανισμός θα ήταν στο ψή, βλέπω να αυξάνονται πολλοί δαπάνες. Και ίσως γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η διασυνοριακές αυτές συνεργασίε να γίνονται επί εθελοντική Γι' αυτό, παραλαμβάνω η δρομολόγηση μέσω Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα έδινε αυτή τη δυνατότητα ακριβώ στα κράτη-μέλη. Και έχουμε μια άλλη νέα πρόταση, τη δυνατότητα μικροχρηματοδότησης κοινωνικών συμπράξεων. Εκπαίδευση για συμβουλευτική καθοδήγηση των ε, δικαιούχων του δικτύου δηλαδή μικροχρηματοδότησης. Πρόκειται για δαπανηρό μέτρο. Βάσει εκτίμησης, που μπορούμε να συζητήσουμε συνεχεία αν θέλετε, για το σύνολο της περίοδου αυτό θα κόστιζε 650.000 ε, σύμφωνα 6.500 ανά δικαιούχο. Αν προηγήσουμε τους δικαιούχους μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια που υπερβαίνει κατά πολύ τον ε, διαθέσιμο προπολογισμό για μικροχρηματοδοτήσει. Και δύο-τρία πράγματα ακόμη, αν μου επιτρέπετε. Το θέμα της διακυβέρνηση, το οποίο δεν προβλεπόταν όντω στο ρελίο Βλέπω εδώ τροπολογίες σχετικά με την διακυβέρνηση για την εισαγωγή κατεξουδότηση πράξεων, συμβουλευτική επιτροπή κλπ. Πώς θα συμβαδίσει όλο αυτό με τους κανόνες της επιτροπολογίας. Γιατί με το Progress είχαμε βρει λύση. Τώρα με τα νέα μέτρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμβατά και επιθυμητά, αν πάση περιπτώσει. Εν τέλει. Και συμπληρωματικότητα με τα άλλα προγράμματα. Ακούστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χρειάζεται όντως η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και με το πρόγραμμα Δίκαιο και Συμμετοχή των Πολιτών κατά των διακρίσεων και ούτω καθεξής. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόγραμμα με αυτόν τον στόχο. Το, θέμα είναι, το ερώτημα μάλλον είναι κατά πόσον η εισαγωγή των μέτρων, η προσθήκη αυτών των μέτρων στο πρόγραμμά μας δημιουργεί επικαλύψεις. Και τέλος, ορισμοί. Η Κομισιόν είχε προτείνει σειρά ορισμών, κάθε φορά που υπάρχει νομική υποχρέωση, για παράδειγμα στις μικροχρηματοδοτήσεις. Δεν ρωτώμεθα λοιπόν αν έπρεπε να δώσουμε επιπλέον ορισμούς. Το ερώτημα είναι εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο προκειμένου και αυτό είναι και το πέμπτο σημείο που μας απασχολεί στο πλαίσιο της εξέτασης των 400 περίπου τροπολογιών που εξετάσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο και θέλω επίσης να πω στον κύριο Ντιό ότι θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή πάλι μαζί σας για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι, <clears throat> ότι έχετε καταλάβει από τις τροπολογίες ότι το Κοινοβούλιο, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας έχουν τις ίδιες ιδέες για μένα, για τις διαμεθοριακές αυτές εταιρικέ σχέσεις, ότι πρέπει να έχουν κάλυψη από ένα οριζόντιο εργαλείο. Πιστεύω ότι επίσης και το πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο για τα προγράμματα αυτά θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που χρειάζεται. Έχω ένα ερώτημα τώρα για το κόστος της ε, πλατφόρμας ίντερνετ για αυτές τις ενέργειες και δεν έχω πάρει κάποια απόφαση. Απάντηση από εσά και πιστεύω ότι και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο EURES. Για τα δικαιώματα συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς απλώς διεκδικούμε αυτά τα οποία μας δίδει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και αυτό είναι μια στάση που υποστηρίζεται από όλες τις ε, πτυχές, από όλες τις παρατάξεις του Κοινοβουλίου. Εγώ υποστηρίζω αυτό το οποίο λέει η Ελιζαμπέθ Σουέντερ. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα για τους δικαιούχους και δεν θα πρέπει να κολλήσουμε στους ορισμούς. Αυτό είναι ένα θέμα φυσικά που συζητούμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Το θέμα δεν είναι να παγιώσουμε αυτούς τους ορισμούς, αλλά θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα να δούμε τα θέματα πιο ευρέως, ακόμα και τα θέματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παραδείγματο η διακίνηση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό έχει χαρακτήρα κοινωνική καινοτομία. Υπάρχουν φυσικά διαφορετικές ερμηνείε, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση και εδώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Μπουλά, ότι δεν πρέπει να έχουμε περιορισμού. Να υπάρχει μια ρευστότητα και δυνατότητα όσμωσης με το κοινωνικό ταμείο, βεβαίως, Υπάρχουν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα για τη χρήση των εργαλείων μικροχρηματοδότησης από την κυρία Κίνγκα Γκέντς. Θέλω γενικά να σας, να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου δώσατε στα θέματα της διαμεθοριακής εταιρική σχέσης και για τις θετικές πτυχές της ε, κινητικότητος δεν πρέπει να το δούμε σε μια αποκλειστική λύση, αλλά είναι μια λύση που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση της ε, ανεργίας των νέων. Δεν αρκεί να πούμε ότι α, ας πηγαίνουν από το ένα μέρος της Ευρώπης στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Αυτό από μόνο του δεν μπορεί να είναι μια οριστική λύση, απλώς θα είναι ένα κομμάτι ενός οπλοστασίου μέτρων για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων αυτών. Θέλω να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο για τη δική της πρόταση. Νομίζω ότι έχω διεξέλθει όλες τις ε, προτάσεις και είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση που θα μας καλύψει όλους. Εξακολουθούν να παραμένουν μικρές εκκρεμότητες, παραδείγματος χάρη για τα ποσοστά χρηματοδότησης, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποθυμίζω λοιπόν, το χρονοδιάγραμμά μας. Ε, οι επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν ε, πρέπει να το πράξουν. Κάποιοι μάλιστα το έκαναν εχθές, ε, κάποιες θα το κάνουν σήμερα και κάποιες τελευταίες αύριο. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις συμβιβαστικέ τροπολογίες στις 20 Ιουνίου για να τις ψηφίσουμε την επομένη. Τέλος πάντων δεν έχουμε και πολλά περιθώρια, αλλά ε, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μίλησα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών για την έκθεσή σας, ώστε οι ιδιαιτερότητες της ε, ε, πρικοδότησης αυτού του προγράμματος ε, να ληφθούν όλος ιδιαίτερος υπόψη, ε, ιδιαίτερα στην ομάδα επαφής με το Συμβούλιο. Φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας για το πρωί. Γύρω από την έκθεση του Τόμας Μαν, επί του οποίου συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Μεταφορών και καλούμαστε να εξετάσουμε στο πλαίσιο μιας ακρόασης τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της Ένωσης και το θέμα της κατάργησης της οδηγίας 96-67. Επειδή βρισκόμαστε σε καθεστώς ενισχυμένη συνεργασίας με την Επιτροπή Μεταφορών, οι ανησυχίες μας ε, βεβαίως πρέπει καταρχάς να αφορούν τις πτυχές της εργασίας, των συνθηκών εργασίας ε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών εδάφους στα αεροδρόμια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οργανώσαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα Πρώτα ε, θα παρέμβει ο ε, εισηγητής μας, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου ζήτησε να παρέμβει και εκείνη συντόμως ε, μέσω του διευθυντή, την Γενική Διευθύνση MOVE, ο Ματιό Μπάλτουιν και μετά θα δώσω το λόγο στους τρεις προσκεκλημένους μας, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα. Έχω ε, λάβει ε, και αιτήματα άλλων ε, συναδέλφων να παρέμβουν στη σημερινή ακρόαση, γιατί ούτως ή άλλως, εγώ το αρνήθηκα γιατί ούτως ή άλλως είχαμε ακούσει την άποψή τους όσον αφορά τα θέματα αυτά στη σχετική ακρόαση που είχε γίνει στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχω λοιπόν δώσει την προτεραιότητα στους τρεις σημερινούς προσκεκλημένους μας έτσι. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή να κάνουμε αυτή την κοινή ακρόαση. Έχουμε τους εμπλεκομένους και έχουμε φυσικά και την εμπειρία των βουλευτών μας που έρχονται από διαφορετικές χώρες. Είναι διαφορετικά τα αεροδρόμια σε μέγεθος στις διάφορες αυτές χώρες, αλλά έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και ως βουλευτές μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα της λειτουργίας των αεροδρομίων. Είναι σημαντικό να έχουμε και μία αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά και να μην είμαστε απλώς μια γνωμοδοτική επιτροπή γιατί τα, εργαζο... τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες για την παροχή υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Έχουμε πάνω χάρη την ε, διακίνηση των ε, βαλιτσών και, του και των εμπορευμάτων, τον ανεφοδιασμό και διάφορα άλλα θέματα. Η Κομισιόν μας έχει τονίσει ότι πρόκειται για ένα συνολικό τζίρο της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν πρόκειται λοιπόν για μικρά ποσά, πρόκειται για ένα σημαντικό οικονομικό τομέα. Υπήρξε μια ε, φιλελευθερωποίηση του τομέα αυτού του 1996 όταν ήμουν εγώ εισηγητής και εξασφαλίσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια φιλελευθερωποίηση και, μια, και ένα άνοιγμα υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτανε ορισμένες προϋποθέσεις. Και ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπήρχε η δυνατότητα να έχουν εργαζομένους υψηλής ποιότητας και οι οποίοι θα είχαν την κατάλληλη αμοιβή. Έχουν φυσικά αυξηθεί από το 1996 τα προβλήματα ως αποτέλεσμα αυτής της υπερβολικής φιλελευθερωποίησης έχουν μειωθεί ιδιαίτερα οι αμοιβέ των εργαζομένων. Δεν έχω λεπτομεριακά στοιχεία εγώ περιμένω ακόμα να έχω τα αποτελέσματα και αυτά τα οποία θα λεχθούν στην ακρόαση αυτή, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η φιλελευθερωποίηση αυτή δεν έχει επιτύχει τον αρχικό στόχο της Κομισιόν να υπάρχει μεγαλύτερη ε, μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Προτείνει τώρα η Κομισιόν να κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες για περαιτέρω φιλελευθερωποίηση να υπάρχουν στα μεγάλα αεροδρόμια και περισσότερες ε, εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα αυτό. Έχουμε κάνει, έχω κάνει πολλές επαφές με πολλούς συνομιλητές οι οποίοι μου τόνισαν ότι αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά μεγαλύτερη πίεση στις εταιρείες θα μειώσει ακόμα τις αποδοχές των εργαζομένων, αυτό σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη που έχουν οι επιβάτες να έχουν εξασφάλιση ότι θα υπάρχει μια ασφαλής μεταφορά τους και δεν είναι προς το συμφέρον γενικά των προτύπων που θέλουμε να εξασφαλίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε όλοι, είναι προς το συμφέρον μας, να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών στα αεροδρόμια και τώρα όλο αυτό είναι υποκίνδυνο. Επίσης η Κομισιόν άφησε να εννοηθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές οφείλεται στις υπηρεσίες εδάφους. Και εδώ θα ήθελα να έχω και καλύτερες απόψεις από τους παριστάμενους στο hearing. Ζήτησα τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων μου και πληροφορήθηκα ε, από τον Επίτροπο Κάλλας για το θέμα αυτό και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι τα οποία προέρχονται από τις υπηρεσίες αυτές εδάφους. Προτείνει η Κομισιόν να υπάρχουν ορισμένε εγγυήσει για την ε, ανάληψη αυτών των υπηρεσιών, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ήδη στην ε, σημερινή συζήτηση. Έχουμε επίσης ε, την ανάγκη να υπάρχουν και διαιτητικές υπηρεσίες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία τίθενται όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μιας εταιρεία και ενός προμηθευτή ή υπεργολάβου. Αλλά υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ επιχειρήσεων, υπάρχει ένας αγώνας για χαμηλότερες τιμές και μια μεγάλη πίεση ανταγωνισμού σε πολλά αεροδρόμια και επομένως είναι μέρος του καθήκον μας να εξασφαλίσουμε όχι μονάχα ότι γίνονται τα πράγματα προς το συμφέρον της αγοράς αλλά και ο καταναλωτής, ο επιβάτης των αεροπορικών γραμμών θα μπορέσει να έχει εξασφάλιση ότι θα διακινείται με ασφάλεια και θα μπορούν να κινούνται όλα τα στοιχεία αυτής της ε, λειτουργίας των αεροδρομίων εμείς λοιπόν ως Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα αυτά μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καλή συνεργασία με τις άλλες ε, ε επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Δίνω το λόγο στον Μάτιο Μπάλτουιν ε, για μια σύντομη παρέμβαση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chairman. I'm very... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος ε, που θα μπορέσω στη γλώσσα του Σέξπιρ και σύντομα όπω είπατε να σα παρουσιάσω την ε, πρότασή μα για τι υπηρεσίε εδάφου. Έχουμε πολύ ρεαλιστικό στόχο με την πρόταση αυτή. Θέλουμε να με βελτιώσουμε τι υπηρεσίε αυτέ και ως προς την αποδοτικότητα και ως προς την ποιότητά τους. Δεν θέλουμε να φέρουμε επανάσταση, θέλουμε απλώς εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα, όπως άλλωστε μόλις επεσήμανε πολύ σωστά ο κύριος Μαν. Θα ήθελα να πω μερικά γενικά πράγματα. Αυτό που προτείνουμε εμείς ε, είναι μία μικρή, μία περιορισμένη αύξηση ανταγωνισμού ε, ως προς τις επιλογές μας, αλλά δεν θέλουμε ε, να υπάρξουν προβλήματα ούτε με την ποιότητα, ούτε με τις συνθήκες απασχόλησης. Και απαντώντας τον κύριο Μάν, θα ήθελα να πω ότι όντως υπάρχουν καθυστερήσεις, ε, όμως ε, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον εγώ δεν λέω, ε, ότι αυτό είναι ευθύνη των εργαζομένων στις υπηρεσίες εδάφους. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτής εξ αρχής. Αυτό που προτείνουμε εμείς σε σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό ως προς την ευρύτερη, τη συνολική ισορροπία ισορροπία της πρότασης Εσείς μιλήσατε για αυξημένο αντιγωνισμό, όμως υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για τις οποίες θα μπορούσε να ήταν πολύ καλή η πρότασή μας για του εργαζόμενους. Πρώτος, ε, πρώτον, ε, η μεταφορά ε, η ισχύουσα οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και επί της βάσης αυτής η Γερμανία και η Ιταλία έδωσαν τη δυνατότητα ε, μετάθεσης των ε, εργαζομένων ε, όταν κάποια υπηρεσία σε κάποιο αεροδρόμιο σταματούσε να λειτουργεί. Υπήρχε όμως μία αμφισημία όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αυτό που προτείνουμε είναι να αποσαφινιστεί αυτό, να δώσουμε τα δικαιώματα στο κράτη, το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να να φροντίσουν το προσωπικό τους σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ε, ε, ε, ενέκρινε την πρόταση αυτή. Η Γερμανία και ε, η Ιταλία αυτή τη στιγμή θα άρχιζε να ισχύει η συγκεκριμένη πρόταση, θα μπορούσε να εφαρμόσει όλα αυτά που αναφέρονται στην πρόταση. Και μπορώ να σα δώσω και ορισμένα παραδείγματα πώ στην πράξη θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, όπω είπατε, σε σχέση με το θέμα αυτό τη εκπαίδευση. Αυτό όμω που θα θέλαμε ήταν να προχωρήσουμε λίγο ακόμη. Κάθε εργαζόμενο που ήδη εκπαιδεύεται τουλάχιστον κάθε δύο, για δύο μέρες το χρόνο ε, να προβαίνει σε μια επιπλέον εκπαίδευση και είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό συνδέεται με το τρίτο σημείο που θέλω να θέσω, ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ελέγχουν ε, τα προσόντα και την ε, εμπειρία των προσωπικών πριν δώσουν την έγκριση, την πιστοποίηση σε μια υπηρεσία ε, σε ένα φορέα εκμετάλλευση ότι ε, μπορεί να αναλάβει τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό είναι για την εξασφάλιση ε, καθαρά τη ποιότητα και των συνθήκων απασχόλησης. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα μέτρα αναφέρονται επαρκώς στην οδηγία. Αντί για, 7, για, αντί για 17 χρόνια ε, ανανέωση των ε, διαγωνισμών, κάτι το οποίο βέβαια έχει άμεση σχέση με την υπεργολαβία. Ε, υπάρχουν επίσης ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας που θέτουν οι αερολιμένες και τα, τα, τα κριτήρια αυτά πρέπει να αναφέρονται ε, στις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Εμείς προσπαθούμε η πρόταση αυτή να παραμείνει ε, λογική και έχουμε αποφύγει όλα τα πολύ ριζοσπαστικά μέτρα ε, για, να, δουν, για, το πλήρες άνοιγμα των υπηρεσιών αυτών Όπω μπορεί να έχουμε κάνει σε άλλου τομεί, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να είχε επιβλαβέ ε, αποτέλεσμα για του εργαζόμενου. Τώρα, για ποιο λόγο η Επιτροπή θεωρεί ότι ε, η κοινωνική πτυχή είναι ένα από, τα βασικά, από τις βασικές παραμέτρους για την υψηλή ποιότητα των ε, υπηρεσιών αυτών, θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στη δική σα υποστήριξη και τη δική σα επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα. Βεβαίω ευχαρίστω να ακούσουμε προτάσεις για βελτίωση του κειμένου και όπως ε, είπατε κι εσείς έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος, υπάρχει κοινό έδαφος πλέον ε, ε, δηλαδή μικρή αύξηση του ανταγωνισμού αλλά ε, με πολύ σημαντικό αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στην ε, ε, αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και πάλι που είναι εδώ σήμερα και προτείνω να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Γιάνντε Λεφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ground Operations των σε Brussels Airlines. Ε, η... Έχετε ε, εμπειρία σε πολλές αεροπορικές εταιρείες και υποθέτω ότι έχετε ε, μια ευρύτερη θεώρηση της κατάστασης και την άποψή σας βεβαίως ήσασταν στη Σαμπένα, στην Air, στην Brussels Airlines και στη Virgin Express. Θα σας δώσω το λόγο για 7 λεπτά και μετά βεβαίως θα μπορείτε να απαντήσετε και στις ερωτήσεις ε, μετά τις παρεμβάσεις των υπολείπων προσκεκλημένων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να καταθέσουμε την υπόψή μας από την άποψη μιας αεροπορικής εταιρεία, της Brussels Airlines, μια σχετικά νέας μικρής εταιρεία που ανήκει όμως στον όμιλο της Lufthansa, δηλαδή της Star Alliance. Brussels Airlines έχει δρομολόγια κυρίως στην Ευρώπη και την Αφρική σε περίπου 3.000 υπαλλήλου. 300 από αυτούς στις Βρυξέλλες, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών ασχολούνται με τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης. Αυτό είναι μια απόφαση που πήραμε, δηλαδή να λάβουμε αυτήν την απόφαση λόγω τη έλλειψη ανταγωνισμού και τη υποβάθμιση των υπηρεσιών προ του επιβάτε. Έχω λοιπόν μια δυναμική ομάδα που απαρτίζεται από νέου ε, εργαζομένου που δουλεύουν στην επίγεια εξυπηρέτηση. Είναι τομέα ο οποίο έχει απελευθερωθεί όπω είναι γνωστό. Τι γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη. Ο τομέα έχει σχεδόν πλήρω απελευθερωθεί. Υπάρχει υπηρεσιών από τους οποίους εξαρτώμεθα για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους επιβάτες μας εν τέλει. Αυτός το μέσο όμως δεν έχει απελευθερωθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν πολλές φορές τριμωγμένοι αν θέλετε και εκεί η αγοραστική μας δύναμη δεν είναι αρκετή. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικέ υπηρεσίε στους πελάτες μας, στου επιβάτε. Αν δούμε λοιπόν τον ευρωπαϊκό χάρτη, όπως είπε και ο κύριος Μάν προηγουμένως, η οδηγία εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και το ξέρουμε αυτό και από τη δική μας εμπειρία. Οι τιμέ, όπως έχουμε δει και αλλού, μειώνονται όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Και όταν όλο αυτό λειτουργεί συντονισμένα, ισορροπημένα, διατηρούμε και την ποιότητα. Πρέπει λοιπόν ο ανταγωνισμός να είναι υγιής, θεμητός, ισορροπημένος για να μπορούμε εν τέλει να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στα αεροδρόμια, στα οποία όπου υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός από άλλα αεροδρόμια. Αν δούμε τώρα την κατάσταση στις Βρυξέλλες, που είναι και η έδρα μας, πολύ σημαντική όπως καταλαβαίνετε για μας, η αγορά δεν έχει πλήρως απελευθερωθεί στον τομέα της διακίνησης των αποσκευών και την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών. Αυτό δυστυχώς, κατά την άποψή μας, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δικαστικές διαμάχες οβούν εδώ και ένα χρόνο περίπου και αυτό δεν βοηθάει την ποιότητα. Όπως είπα, υπάρχει αδιέξοδο για τις αεροπορικές εταιρείε, για τους επιβάτες και σίγουρα για τους υπαλλήλου τόσο των αεροπορικών εταιριών όσο και των εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης. Όλα αυτά εν τέλει θα είναι κατά των υπαλλήλων και θα δημιουργηθεί φοβούμε χάος όταν η αγορά απελευθερωθεί με ασαφείς όμως κανόνες. Θα μπορούσε η απελευθέρωση μάλιστα να οδηγήσει σε ιονή μονοπόλια, διότι οι δύο πάροχοι επιγείες εξυπηρέτηση που πήραν πριν από ένα χρόνο περίπου τη σχετική άδεια, είπαν ότι ο ένας πάροχος θα απορροφηθεί από τον άλλον. Άρα μιλάμε για δύο άδειε οι οποίε εν τέλει θα ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Η πρόταση της Κομισιόν που προβλέπει τρεις εταιρείε και όχι δύο για αεροδρόμια με πάνω από 5 εκατομμύρια επιβάτε είναι μια καλή πρόταση. Βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και την υποστηρίζουμε. Πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία οι τελικοί χρήστες οι αεροπορικές εταιρείε πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν καλές υπηρεσίες στους τελικούς αποδέκτες, τους επιβάτες. Και έτσι πρέπει να δούμε τις υπηρεσίες παροχής επιγής εξυπηρέτησης στα διάφορα δρόμια. Ας δούμε τώρα τα επιμέρους στοιχεία της ε, σημερινής πρότασης. Η Brussels υποστηρίζει εν γέννη την πρόταση της Κομισιόν, όμως χρειάζεται προσοχή και σύνεση. Εμείς δεν θέλουμε οποιοδήποτε να πηγαίνει σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο και να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία. Όχι, θέλουμε ένα προσεκτικό, λελογισμένο άνοιγμα της αγοράς που θα δώσει την δυνατότητα σε περισσότερες εταιρείε που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους και τη φροντίδα για τους υπαλλήλους να μπουν πιο εύκολα όντως σε περισσότερα αεροδρόμια. Αυτό για μας είναι ένα στοιχείο κλειδί για να βελτιωθεί η υπηρεσία που εν τέλει παρέχουμε προς τους επιβάτες. Και μιλώ για την ακρίβεια των πτήσεων, τις αποσκευές, τον εφοδιασμό κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καθυστέρηση μιας πτήσης δεν είναι θέμα, δεν είναι ευθύνη ενό εργαζομένου, αλλά του συστήματο γενικότερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν υγιή ανταγωνισμό και αυτό θα επηρεάσει και το θέμα του κόστους. Για να σας δώσω και μερικά νούμερα ε, σε εμά και φυσικά αυτό διαφέρει από εταιρεία σε αεροπορική περίπου 15% του συνολικού κόστους μας αφορά την επίγεια εξυπηρέτηση. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίε πηγέ εξυπηρέτηση, οτιδήποτε συμβαίνει στο έδαφο. Αυτό σα δίνει λοιπόν μια τάξη μεγέθου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να μειώσουμε τι τιμέ μα περαιτέρω, χρειαζόμαστε και τη σχετική απελευθέρωση με προσοχή και σύνεση, όπω είπα όμω, από ανθρώπου και εταιρείε που έχουν αποδείξει την αξία του και την ικανότητά του, χωρί να διακυβευτεί βεβαίω και η ασφάλεια. Προσωπικό. Πιστεύουμε ότι και εδώ πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και προστασίας των εργαζομένων. Να παραμείνουμε λοιπόν ανταγωνιστικοί. Ε, μετά έχουμε τις εθνικές ιδιομορφίες, την εθνική νομοθεσία, την προστασία της εργασίας και εν τέλει η προστασία της τεχνολογίας που διαθέτει το προσωπικό. Οι εταιρείε που παρέχουν πηγή εξυπηρέτηση πρέπει να επιλέγουν τους εργαζομένου, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο για να μπορούν να παρέχουν και τις απαραίτητες υπηρεσίες, τις ποιοτικέ υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται λοιπόν για μείωση αυτών των μισθών. Πολλές φορές μάλιστα το έμεσο κόστος είναι υψηλότερο. Μιλάμε λοιπόν για ένα ε, σύστημα, αλλά και για του υπαλλήλου που εν τέλει παρέχουν την υπηρεσία και που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο ανταγωνισμό σε κάθε περίπτωση πάντω πρέπει να ανοίξει προσεκτικά. Η ποιότητα είναι πολύ σημαντική. Επίση υπάρχουν ένα σωρό κανονισμοί αυτή τη στιγμή. Ω αεροπορική εταιρεία εμεί είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια κατά γνώμων ενεργειών και ατυχημάτων για του επιβάτε. Τελικά. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ΑΙΑΤΑ, ΑΙΣΑΓΟ και άλλων διεθνών οργανισμών. Έχουμε ενσωματώσει τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει λόγος να περιγράψουμε με την τελευταία λεπτομέρεια τις ποιοτικέ απαιτήσει, διότι διαφέρουν εν γέννη από αγορά σε αγορά, από χώρα σε χώρα, από κατάσταση σε κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτές, Ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα της κατάστασης όπως τη βλέπουμε εμείς ως Brussels Airlines τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στον επόμενο. Το μιλτή μας, τον κύριο Ιγκο Φουσφος, εκπροσωπεί τους εργαζομένους ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΟΥ ΑΖΕ. Ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε βέβαια καλύτερα εσείς ποιους ακριβώς εκπροσωπείτε και τι σημαίνει το ακρόνιμο αυτό και να μας παρουσιάσετε φυσικά και τη θέση σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ja, herzlichen Dank. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Μπέρες, τον κύριο Μαν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας για την διενέργεια αυτής της ακρόασης και για το γεγονός ότι γίνεται ακουστή και η άποψη των εργαζομένων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της σημασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι θετικό στοιχείο για τον κοινοβουλευτισμό ότι μπορεί να ακούει αντιμαχόμενες απόψεις αυτά τα θέματα οι, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ε, ξέρουν ότι σε πολλές άλλες ε, ακροάσεις δεν ακούγονται καθόλου οι απόψεις των συνδικάτων και τους αφήνουν έξω από την πόρτα. Η, τα συνδικάτα λοιπόν για τις μεταφορές στη Γερμανία είναι αυτά τα οποία καλύπτουν την, ε, τις υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια αλλά σήμερα είναι και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που έχουν υπό την αιγύδα τους 85 συνδικάτα που είναι δραστήρια στα θέματα των υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνουμε όχι μονάχα αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τις υπηρεσίες εδάφους, αλλά και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με άλλες υπηρεσίες όπως είναι η κατεύθυνση των αεροπλάνων στο, στα αεροδρόμια, υπηρεσίες τροφοδοσίας κτλ. Δεν είμαστε λοιπόν μια μικρή μονάχα ε, ένα μικρό συνδικάτο, αλλά εκπροσωπούμε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων στα αεροδρόμια. Η εντύπωσή μας είναι ότι η Κομισιόν σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία δεν έχει σκεφτεί καλά και δεν έχει επεξεργαστεί την ε, πρότασή της. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι η πρόταση της Κομισιόν θα καλύψει τις ανάγκες αυτών των ατόμων που εργάζονται στην εξυπηρέτηση εδάφου. Λέει η Κομισιόν ότι είναι 60.000 στην Ευρώπη, αλλά μόνο στη Γερμανία είναι 40.000 αυτοί που εργάζονται στην εξυπηρέτηση εδάφου. Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 300.000 όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στην εξυπηρέτηση εδάφους και οι οποίοι πρέπει να καλυφθούν από αυτή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μονάχα τα άτομα αυτά τα οποία είναι σε άμεση σύνδεση με, την εξυπηρέτηση εδάφου, Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι <clears throat> είναι εργαζόμενοι όπως είναι και οι πιλότοι και το άλλο προσωπικό των αεροπορικών εταιριών που εμπλέκονται γενικά σε αυτήν την εργασία και πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ότι οι βαλίτσες των επιβατών θα έρθουν στην κατάλληλη στιγμή και ότι υπάρχει η απαραίτητη κατάρτιση των ε, πληρωμάτων και των εξυπηρετητών των αεροσκαφών ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλεία τους. Επομένως είναι θέματα που ξεπερνούν απλώς τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες εδάφους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ευρύτερες, είναι οριζόντιες. Έχουμε γενικά να αντιμετωπίσουμε από την Πορτογαλία ως την Πολωνία επισφαλής ε, συνθήκες εργασίας. Έχουμε άτομα τα οποία έχουν μονάχα μερικέ ώρες εγγυημένη εργασίας το μήνα και τους καλούν την τελευταία στιγμή για να, να έχουν ένα μεροκάματο παραπάνω. Έχουμε άτομα λοιπόν τα οποία εργάζονται σε συνθήκες οι οποίες είναι επισφαλείς και για όλες τις χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτός ο αποσπασματικός τρόπος εργασίας αλλά ιδίω σε χώρες οι οποίες έχουν απορρίθμιση της αγοράς. Στη, χώρα που γνωρίζω πολύ καλύτερα από τις άλλες είναι ότι μετά από τη θέση εφαρμογή της τωρινής οδηγίας 40% των ε, εργαζομένων στην εξυπηρέτηση εδάφους πληρώνονται με την ώρα και δεν τους φτάνει καν αυτό το εισόδημα που έχουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. 20% <clears throat> και πάνω των θέσεων εργασίας έχουν υποστεί πραγματική διάβρωση της, ε, των αποδοχών τους. Υπήρξε απώλεια θέσεων απασχόλησης επίσης. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες <clears throat> αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση εδάφους και αμέσως απολύουν σχεδόν το μισό του προσωπικού. Είδαμε να έχουμε εμπειρίες αυτού του είδους ότι ενώ στο παρελθόν υπήρχε μια σωστή κατάρτιση για την εξυπηρέτηση εδάφους και η οποία χρειαζόταν μήνες για να συμπληρωθεί υπάρχουν τώρα εταιρείες οι οποίες δεν κάνουν καν κατάρτιση των εργαζομένων τους. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα αυτό και αναφέρονται κάποια από αυτά τα προβλήματα στο έγγραφο της Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι ότι οι προτάσεις που κάνει στη συνέχεια η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα δεν είναι ορθές, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αν εφαρμοστεί η πρόταση της Κομισιόν στις χώρες όπου μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά, εκεί η κατάσταση σταδιακά θα γίνει ακόμα χειρότερη, θα μειωθεί η ποιότητα εξυπηρέτηση και θα χάσουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι τις θέσει εργασία τους. <clears throat> Ενώ στι χώρες όπου η κατάσταση είναι ήδη ε, αρνητική, εκεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερες επιδενώσεις. Γι' αυτό και κλείνω, έχουμε πέντε κύριες διεκδικήσεις ως ε, συνδικάτα εργαζομένων στον αεροπορικό τομέα. Πρώτα απ' όλα δεν θέλουμε να υπάρξει καμία διεύρυνση της υποχρεωτικής επιβολής ε, εταιριών για την εξυπηρέτηση εδάφους χωρίς να τροποποιηθούν οι συνθήκες εργασίας. Δεύτερη αίτηση, να αποφευχθεί να υπάρξει ανταγωνισμός που οδηγεί σε μισθολογικό ντάμπινγκ. Βεβαίως να υπάρχει ανταγωνισμός σε σχέση με την καλύτερη ποιότητα, αλλά όχι προς την κατεύθυνση του ντάμπινγκ. Το άρθρο 98 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να απαγορεύσει οι εταιρείε αυτές να κάνουν ουσιαστικά μια εικονική μορφή ανταγωνισμού για να διώξουν τις πιο σοβαρές εταιρείε από τον τομέα αυτό. Επίσης αυτό σημαίνει ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να εξασφαλίζουν για τα αεροδρόμια τους ότι οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες έχουν συναυθεί εφαρμόζονται πράγματα. Τρίτον, όταν υπάρχει αλλαγή υπηρεσίες θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να μεταφερθούν στη νέα ε, επιχείρηση που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση εδάφους χωρίς μισθολογική ε, απώλεια. Η Κομισιόν αυτό το θέμα το έχει θέσει μονάχα προαιρετικά και δεν είναι τυχαίο ότι η Κομισιόν έχει βρεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λόγω αυτής της ε, θέσης. Τέταρτον, θέλουμε να υπάρχει μια μόνιμη παραχώρηση υπεργολαβίας σε άλλες εταιρείες. Ξέρουμε ότι σε προσωρινό επίπεδο μπορεί να είναι κάτι το απαραίτητο, αλλά η εμπειρία μας με τις υπεργολοβίες είναι ότι η εταιρεία παίρνει, μια εταιρεία παίρνει μια άδεια για την εξυπηρέτηση εδάφους και μετά τα δίδει αυτά τα δικαιώματα με υπεργολαβία σε μια εταιρεία η οποία δεν πλήρει τις προδιαγραφές για μια α, ποιότητα εξυπηρέτησης. Η πέμπτη και τελευταία βαστή εκδίκηση είναι ότι θα θέλαμε να υπάρξουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα αυτό και επίσης να υπάρχει μια ανάγκη για να γίνονται θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σε σχέση με την ικανότητα των ατόμων αυτών. Όταν λέει η Κομισιόν ότι για κάθε συγκεκριμένο τμήμα των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να κάνουν μονάχα δύο μέρες ε, κατάρτιση εργαζόμενων. Εγώ δεν θέλω να με ένα αεροπλάνο που οι φορτωτέ του έχουν περάσει μονάχα μια εκπαίδευση δύο ημερών. Με τις προτάσεις αυτές εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Η ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνική και η Οικονομική Επιτροπή έχει ζητήσει και αυτή στη γνωμοδότησή της να υπάρξει μια επανεξέταση των θεμάτων αυτών και τα κύρια αυτά σημεία τα οποία έχουμε αναφέρει ως συνδικάτα τα έχουν αποδεχθεί. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ αν εσείς ως μέλη της ε, Επιτροπής Απασχόλησης σκεφτείτε καλύτερα για αυτές τις απόψεις και ενδεχομένως δεχτείτε κάποιες από αυτές τις διεκδικήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Donc nous... Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην, στον τελευταίο μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κριστόφ Κέψεν, ε, που είναι Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων ε, στην ACI Europe. Ε, διεθνές, το Διεθνές Συμβούλιο δηλαδή αερολιμένων και θα μας παρουσιάσετε τις δομές των αεροδρομίων. Στο παρελθόν έχετε εργαστεί και στο... Ε, ε, ορικό επιμελητήριο Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε ε, και και έχετε κάνει και σπουδές στην Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή σας που μας κάλεσε εδώ σήμερα για να σας πούμε την άποψή μας όσον αφορά τις κοινωνικές πτυχές ε, του ε, κανονισμού για τις υπηρεσίες εδάφους. Πριν πω σε λεπτομέρειες για τον προτινόμενο ε, κανονισμό, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τον οργανισμό που εκπροσωπώ. Εμείς έχουμε την έδρα μας εδώ στις Βρυξέλλες, εκπροσωπούμε περίπου 400 αεροδρόμια ε, ευρωπαϊκά και επίσης ε, η συνέτεροι μας ε, είναι οργανώσεις αεροδρομίων όπως επίσης και εταιρείες υπηρεσιών εδάφους το βασικό σημείο εστίγασης ε, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών εντάφους. Αν δει κανείς τι σημαίνει κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως αναφέρθηκε κάτι τέτοιο στις προηγούμενες ε, ε, παρεμβάσεις, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, η τροφοδοσία, η συντηρήση του αεροσκάφους, ο καθαρισμός, ε, ε, υπηρεσίε φορτίου και ταχυδρομείου, μεταχείριση ε, επιβατών και αποσκευών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα στα αεροδρόμια και παράλληλα να παραμένουν σε μια υψηλή ποιότητα. Ε, υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ των ε, ε, αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ αποτελεσματικές υπηρεσίες εδάφους στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουμε τις περισσότερες κατηγορίες ε, ήδη απελευθερώσει και ορισμένες είναι πολύ πιο περιορισμένες ε, με ελάχιστο αριθμό ε, αδειών. Θα ήθελα απλώς να πω ορισμένα πράγματα για τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, γιατί αυτό δεν το αναφέραμε. Πολλές φορές ε, μιλάμε για λόγους χώρου, ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος ε, για ε, τις υπηρεσίες εδάφους. Μιλάμε για την αποτελεσματικότητα επίσης, γιατί πολλές φορές ο όγκος της κυκλοφορίας είναι ε, πολύ χαμηλός ε, για να υπάρχουν ε, πολλές, πολλοί φορείς και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα υπήρχε ακόμη υψηλότερη πίεση για τομείς όπως οι τιμές και οι κοινωνικές συνθήκες και υπάρχουν επίσης και τα ζητήματα ασφαλείας. Όλο και περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης ε, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερος, υπάρχουν και μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Σήμερα η αγορά, στην αγορά επικρατούν οι ανεξάρτητες υπηρεσίες εδάφους. Αν δείτε τα νούμερα θα δείτε ότι το 1996 όταν ε, εγκρίθηκε η πρώτη οδηγία οι αεροπορικές εταιρείες ε, επικρατούσαν, έχει αλλάξει το 2010, έχουν αντιστραφεί τα ποσοστά. Πρώτη είναι οι ανεξάρτητοι φορείς και μετά είναι οι αεροπορικές εταιρείες ε, και οι ε, φορεί διαχείριση των αεροδρομίων έρχονται τελευταίε με 16%. Τώρα, πρέπει να μιλήσουμε ειδικότερα όσον αφορά τις πτυχές της εργασίας ε, για την τρέχουσα κατάσταση. Ε, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου της Επιτροπής, 65 με 80% του κόστους υπηρεσιών εδάφους ε, ε, έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Αν λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά, συμβαίνει ότι υπάρχει, συνήθως το αποτέλεσμα είναι και ανταγωνισμός στις τιμές. Αν 65 με 80% του κόστους αφορούν το προσωπικό, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι υπάρχει πίεση όσον αφορά τις κοινωνικές συνθήκες, ε, για το προσωπικό και ειδικότερα για τους μισθούς. Ε, αναφέρθηκαν άλλωστε και τα στοιχεία τα σχετικά από, τους, ε, από τα συνδικάτα. Έχουμε δει μειώσεις των μισθών σε κάποιες χώρες και επίσης έχουμε δει και μείωση των τιμών στην αγορά αυτή. Από το 1996 υπήρξε μια αύξηση περίπου 25% των τιμών, των τιμών υπηρεσιών εδάφους, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια κατάσταση ε, πολύ μικρών περιθωρίων όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές, όμως ένα ε, περιβάλλον μεγάλου ανταγωνισμού. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη πίεση ε, και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων αλλά και για την ποιότητα των αεροδρομίων. Μία από τις συνέπειες που προέκυψαν είναι ότι, είναι ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, οι αεροπορικές εταιρείες, ε, τα συνδικάτα, οι ανεξαρτητε φορείς ε, υπηρεσιών εδάφους και Υπήρξε μια κοινή δήλωση με, εκ μέρους των τριών από τους τέσσερις κοινού, ε, κοινωνικούς εταίρους. συμφώνησαν σε ένα σύνολο μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν όταν θα αναθεωρηθεί η οδηγία και για τις κοινωνικές ρήτρε και για τη διαδικασία των διαγωνισμών και υπήρξαν και κάποια γενικά σχόλια όσον αφορά την περαιτέρω απελευθέρωση της ε, ε, αγοράς αυτής και τα ενδεχόμενα προβλήματα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας την υπέβαλε το Δεκέμβριο του 2011 λέει ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω απελευθέρωση με ελάχιστο, ε, με ελάχιστο, ελάχιστη αναφορά πέντε αεροδρόμια, ε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κατά τη γνώμη μας σημαίνει πίεση για τις τιμές και για τις ε, συνθήκες εργασίας και γι' αυτό αμφισβητούμε αυτή τη δογματική προσέγγιση για το περαιτέρω άνοιγμα των υπηρεσιών αυτών. Η απελευθέρωση δεν είναι ε, κατά τη γνώμη μας ε, ε, μια πολύ γενική προσέγγιση που τα είπε η Πισοπεδόνδη Διόλα. Πρέπει να δούμε και τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν. Είδαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, ότι η εισηγήτρια της Επιτροπής Μεταφορών, ο εισηγητής, συγγνώμη, υπέβαλε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις και ακόμη αναλύουμε τις προτάσεις αυτές. Βλέπουμε όμως ότι προτείνει να πάμε πέρα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τέσσερις ε, διαγωνισμούς στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και να αλλάξουμε και τον ορισμό μάλιστα της ε, έννοιας της εξυπηρέτησης εδάφους με ίδια μέσα από τα αεροδρόμια. Αυτά κάπως μας ανησυχούν. Όσον αφορά τώρα τις κοινωνικές ε, εγγυήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ε, πολύ καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση, όμως θα θέλαμε να υπάρχει μια δεσμευτική μετάθεση των, ε, του προσωπικού, κάτι το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 12. Δεν θα θέλαμε σε εθνικό επίπεδο να γίνουν τεράστιες συζητήσεις κατά πόσο θα έπρεπε να, να εφαρμοστούν σχετικοί νόμοι, να εγκριθούν σχετικοί νόμοι για τη μετάθεση των εργαζομένων. Θα θέλαμε να υπάρχει ένα δεσμευτικό άρθρο και μιλάω για το άρθρο 12 ως προς το θέμα αυτό. Οι, απαιτήσεις, οι ελάχιστες απαιτήσει ε, εκπαίδευσης δύο ημερών ε, είναι μία πρόοδο σε σχέση με την ισχύουσα οδηγία, αλλά δεν είναι παρκές. Εμείς θα προτιμούσαμε μία εβδομάδα, γιατί αυτό είναι ο χρόνος που χρειάζεται ε, για την εκπαίδευση σε, σε αιτήσια βάση, όμως βεβαίως συζητήσιμο είναι αυτό και ευχαρίστως να το συζητήσουμε στην Επιτροπή σας. Αλλά βασική βασικοί τομείς ε, είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές, οι ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας. Για μας αυτό είναι σημαντικό. Ε, πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να γίνονται σεβαστές ε, από όλους τους ε, φορείς που δραστηριοποιούνται σε ένα αεροδρόμιο. Συνήθως βέβαια η σύμβαση είναι μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του φορέα παροχής της υπηρεσίας. Εμείς δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει μια ελάχιστη ποιότητα την οποία να σέβονται όλοι ότι ε, οι υπηρεσίες γενικώ στο αεροδρόμιο λειτουργούν εύρυθμα και να μην φτάνουμε σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει, πολύ, υπάρχει κακή ποιότητα λόγω κακής επίδοσης κάποιων μεμονωμένων φορέων. Υπάρχουν κάποιες ακόμη διατάξεις που κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικές για τα αεροδρόμια, όπως για παράδειγμα η Κομισιόν αναφέρεται ε, σε νομικό διαχωρισμό μεταξύ ε, των ε, φορέων εκμετάλλευσης και της κάποιες πιο κεντρικής δομής. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά για μας είναι πάρα πολύ προβληματικό αυτό το θέμα. Είναι κάτι που δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις υπηρεσίες εδάφους και θα θέλαμε να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν ισότιμοι ε, όροι. Γι' αυτό ε, δεν συμφωνούμε με αυτόν τον νομικό διαχωρισμό. Και υπάρχουν επίσης και κάποια ζητήματα για το διοικητικό φόρτο, κάποιες διτάξεις του διοικητικό φόρτο που θα πρέπει να βαρύνει και τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και τους αερολιμένες σε σχέση με κάποιες πιο κεντρικές δομές. Εμείς θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε αυτή την πρόταση με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η κατάλληλη. Ε, θα ήθελα να ολοκληρώσω ανακεφαλαιώνοντας τις ε, προτεραιότητές μας. Ε, για μας το σημαντικότερο θέμα είναι η ποιότητα πρέπει να έχουμε τα εργαλεία για να θέτουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές σε ένα αεροδρόμιο. Δεν θέλουμε δογματική προσέγγιση για την ε, απελευθέρωση, να διατηρήσουμε μεν τις διατάξεις, αλλά να αφήσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν αν θα απελευθερώσουν την αγορά ή όχι. Θέλουμε περισσότερες κοινωνικές ε, ρήτρε, ε, δεσμευτικό άρθρο 12 και αυξημένη εκπαίδευση για το προσωπικό εδάφους. Επίσης ε, θα μας ικανοποιούσε ιδιαίτερα εάν η άποψη των κοινωνικών εταίρων, των συνδικάτων και των ανεξάρτητων ε, της, ε, που ανέφερα άλλωστε την κοινή τους δήλωση θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της γνωμοδότησης για τον κανονισμό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μας μένει μισή ώρα και κάτι για συζήτηση. Ποιος θέλει τον λόγο, και μετά κυρία Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή. Είναι και η ελπίδα μου ότι η έκθεσή του θα πάει προς την κατεύθυνση που η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να κατανοηθεί καταρχήν ότι δεν έχουμε μονάχα ένα καθαρά γερμανικό πρόβλημα. Τα προηγούμενα ε, χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχες κατάστασεις υπερφιλελευθεροποίησης, παραδείγματος χαρή ο τομέας των ταχυδρομείων, που οδήγησαν σε μία μείωση της ποιότητας για τον καταναλωτή, αλλά και φυσικά και σε μία επιδείνωση των συνδικών εργασίας <clears throat> για τους εργαζομένους. Και αν δω λοιπόν πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά από τις πρώτες προσπάθειες φιλελευθεροποίησης. Είναι εύγλωτα τα στοιχεία, υπάρχει σημαντική αύξηση στις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μείωση των ε, αποδοχών και μείωση των επενδύσεων σε κατάρτιση των εργαζομένων. Και όταν πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι οι υπηρεσίες στον αεροπορικό τομέα και όπου υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες αυτού του είδους. <clears throat> Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη την κοινή θέση των Ευρωπαίων <clears throat> κοινωνικών εταίρων. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν γίνει σαφή από αυτή τη γνωμοδότηση. Και έχω να θέσω τρία ερωτήματα προς τους ομιλητές που έλαβαν τον λόγο προηγουμένως. για τον εκπρόσωπο της Brussels Airlines. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πράγματι πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός σημαίνει χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάτω από το 1% η συμμετοχή τη εξυπηρέτηση εξυπηρέτησης στο συνολικό κόστος των αεροπορικών ναύλων. Και επομένως είναι αυτό κάτι το οποίο κάνει τόσο απαραίτητη την ε, φιλελευθερωποίηση. Εγώ πήγα πρόσφατα στη, στην ε, Αραβική Χερσόνησο και είδα ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στο Αμπού Ντάμπι και στο Ντουμπάι κτλ. Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να είσαστε ανταγωνιστικοί όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες εργασίας. και πώς ε, θεωρείται ότι πρέπει να εξελιχθεί ο ανταγωνισμός. Στον εκπρόσωπο της Βέρντι τώρα, του Συνδικάτου των ε, Εργαζομένων στον τομέα αυτό, μιλήσατε για τις εξελίξεις των τελευταίων δέκα ετών. Υπάρχουν τώρα κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αν υπάρξει μια πλήρης εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Πώς έχει η κατάσταση επίσης για τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας, πώς έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. <clears throat> και για τον εκπρόσωπο των αεροδρομίων, ποιες είναι οι ανησυχίες ασφάλειας που υπάρχουν από την πλευρά των αεροδρομίων σε σχέση με, τους, ε, με τις εταιρείες ε, που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση εδάφους ποιες είναι οι απαιτήσει ασφαλείας που θα πρέπει να εκπληρούνται από τις ε, ε, εταιρείε αυτές και αν αυτό θα γίνει προβληματικό με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Θέλω να περιοριστώ λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία μονάχα. Ναι, γερμανικό το πρόβλημα. Δίνω το λόγο όμω στην κυρία Ήρς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αναφέρεται πάντα το θέμα της φιλελευθερωποίησης και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ως εκπρόσωπος των φιλελευθέρων θα πετάω από τη χαρά μου. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα είναι απαραίτητο να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Aber, ähm, ich denke auch, dass man... Äh, Μιλάμε λοιπόν για την ποιότητα των υπηρεσιών κυρίω. Ξέρουμε ότι ήδη και τώρα έχουμε μία μορφή ένα ανταγωνισμό. Πολλά αεροδρόμια έχουν πράγματι παραπάνω από ένα πάροχο υπηρεσιών στον τομέα αυτό. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι το πιστεύουν ότι είναι καλύτερος ο ανταγωνισμός, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το παράγοντα κόστος αλλά και τον παράγοντα ποιότητος. Ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια πίεση ε, κόστους και φυσικά είναι γνωστό αυτό και ότι αντιμετωπίζουν και τον ανταγωνισμό από τις εταιρείε από τον αραβικό από την Αραβική Χερσόνησο. Ξέρουμε επίσης ότι η εξυπηρέτηση εδάφους είναι ένταση εργασίας. Επομένως το προσωπικό είναι αυτό που βρίσκεται στο κέντρο αυτών των ε, ε, υπηρεσιών και το μισθολογικό του κόστος παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Αν λοιπόν η φιλελευθοποίηση για μένα σημαίνει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι θα μειωθούν δραστικά οι αποδοχές των εργαζομένων και τελικά θα πρέπει να καλύπτει το κενό το κράτος με επιδόματα και πρόσθετες, ε, πρόσθετο κόστος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημα μιας τέτοιας ενέργειας να φέρνουμε την αγορά σε μια κατάσταση όπου τελικά το κράτος θα πρέπει να επανέλθει για να καλύψει, για να πληρώσει τα σπασμένα ουσιαστικά. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή τη λειτουργία της απελευθέρωσης πώς την αντιμετωπίζετε. Είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης, επομένως μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το άρθρο 6 και το ερώτημα είναι κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να το εφαρμόσουμε αυτό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι τα προβλήματα τα μισθολογικά. Κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι το θέμα των υπεργολαβιών. Μάλλον, συγγνώμη, το πρόβλημα της ε, τη δυνατότητα να μεταφέρεται το προσωπικό από μια εταιρεία σε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την ε, ε, υπηρεσία αυτή. Δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως μια ε, ασφάλεια γιατί μπορεί τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα να περάσουν στην επόμενη εταιρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να απολυθούν αμέσως στη συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και το ερώτημά μου προ του ομιλητέ είναι πώ αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα τη δυνατότητα μεταφορά των εργαζομένων. Επίση, για το θέμα τη περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε αυτό προ το συμφέρον των εργαζομένων, αλλά αυτό είναι και κάτι το οποίο βρίσκεται προ το συμφέρον των επιβατών. Πιστεύω ότι και οι επιχειρήσει, οι αεροπορικέ επιχειρήσει έχουν κάθε συμφέρον ότι όσο φθηνέ και να είναι οι ενέργειες εξυπηρετήσει θα πρέπει να είναι αποτελεσματικέ έχω πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη όλες αυτές οι προτάσεις της Κομισιόν. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και μια έκθεση αντικτύπου από την πλευρά της Κομισιόν να ξέρουμε πού θα προκύψει κόστος και ποιος θα το επομιστεί και ποιες θα είναι οι συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν από αυτές τις ενέργειες. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να ξέρουμε ότι το κόστος θα προκύψει για το α ή το β κράτος μέλος όταν έχουμε λοιπόν τι προτάσει τη Κομισιόν, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε ποιε είναι οι επιπτώσει και μέχρι στιγμή από αυτά που έχει, έχω δει από την πρόταση τη Κομισιόν δεν ξέρω πώ θα εκτιμήσω αυτέ τι συνέπειε. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα στου τρει ομιλητέ. Πώ αξιολογείται λοιπόν τον αντίκτυπο που θα προκύψει από αυτά τα μέτρα τη Κομισιόν. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Το Χέντερ και Λοιπόν, δεν πρέπει εδώ να τα δούμε τα θέματα αυτά με τα, τις παροπίδες του φιλελευθερισμού. Να λέμε ότι πρέπει να αφήσετε ελεύθερη την αγορά και μετά βλέπουμε ότι το κράτος αναγκάζεται να επανέλθει. Η φιλελευθερωποίηση αυτή, όπως τη βλέπει η Κομισιόν, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στις υπηρεσίες εδάφους οι οποίες από κοινωνική άποψη δεν μπορεί κανείς να την υπερασπιστεί και σε επίπεδο ασφαλείας γίνεται σχεδόν απαράδεκτη για τους καταναλωτές, για τους χρήστες των αεροπορικών εταιριών. Η υπερφιλελευθερωποίηση της Κομισιόν σημαίνει ότι έχουμε 40% περισσότερου εργαζομένου, οι οποίοι όμω πρέπει να ξεπηρετήσουν 100% περισσότερε πτήσει. Και επίσης η μείωση των ε, αποδοχών λόγω του dumping αυτού και τη οργανωμένης απορρίθμιση που έχει προωθήσει η Κομισιόν έχουμε 20% λιγότερες αποδοχές των εργαζομένων στην εξυπηρέτηση εδάφου. 40% από τα άτομα αυτά βρίσκονται στο κατόφλι τη ένδυας. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος φιλελευθεροποίησης λοιπόν. Αυτή είναι μια νοοτροπία λοιπόν η οποία πρέπει να αλλάξει άρδιν. Δεν, δεν θέλω να διαμφισβητήσω την έννοια της ε, φιλανθρωπήσει. Θα μπορούσε να έχει 60 παρόχου υπηρεσιών το κάθε αεροδρόμιο. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν οι συνθήκες ασφάλειας και οι συνθήκες κοινωνικής προστασίας για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Αυτό είναι κάτι που θα το, πρέπει να το δει το κάθε αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση στον τομέα της εξυπηρέτησης εδάφους και να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με έναν τρόπο ο οποίος είναι αποτρόπαιος από πλευρά εργασιακή, κοινωνική και ακόμα και από, πλευρά, από πλευράς ασφαλείας. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν συστήματα τα οποία ουσιαστικά στέλνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους στο περιθώριο. Θέλω να θέσω τώρα τρία ερωτήματα. Πρώτον, είναι σωστό αυτό που είπε ο εκπρόσωπος των αεροδρομίων ότι δεν ε, καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου οι, οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρέτησης εδάφους. Επίσης, και αυτό το οποίο ανέφεραν και οι εκπρόσωποι της ε, Brussels Airlines ότι ουσιαστικά με την φιλελευθερωποίηση μπορεί να κερδίσουμε 1,6 ευρώ σε ένα εισιτήριο 200 ευρώ. Αυτό είναι πραγματικά γελίο μας σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αυτό με την ε, ε, ενώπιον των κοινωνικών συνεπειών που προκύπτουν. Αυτό πρέπει να είναι τελείως αμεληταίο στοιχείο του ανταγωνισμού. Χρειάζεται η Κομισιόν για να κερδίσει αυτό το 1,60 ευρώ να φέρει στο επίπεδο της αθλειότητας του εργαζομένους. Και τρίτον το ερώτημα αυτό που θέλω να θέσω είναι αν είναι γεγονός ότι σε εν μέρη στα γερμανικά αεροδρόμια υπάρχει μονάχα ένας ο οποίος είναι ειδικευμένο στα θέματα αυτά και είναι υπεύθυνο για τρία αεροπλάνα συγχρόνως και πρέπει να ελέγχει τα άτομα τα οποία εξυπηρετούν αυτά τα αεροπλάνα και που ενδεχομένως δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένα εγώ σαν επιβάτης πρέπει να νιώθω μεγάλη ανησυχία για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να έχω τις θέσεις σας για το πώς θα ε, εξασφαλιστεί η ασφάλεια κάτω από τέτοιες συνθήκες στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Ευχαριστώ. Μπέκερ, καταρχήν και μετά να κλείσουμε. Θα πρέπει να ε, αποδεχθείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στα θέματα αυτά. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για την έννοια της φιλελευθεροποίησης. Δεν έχω δει κάποια επιχειρήματα τα οποία να είναι πιστικά, τα οποία να μπορέσουν να εξηγήσουν γιατί κάνουμε αυτή τη φιλελευθεροποίηση σε βάρος των εργαζομένων. Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας εδώ. Στους τομείς αυτούς που και με αυτά τα οποία βλέπουμε βλέπουμε ότι η μία φιλελευθερωποίηση η οποία αφορά το μισθολογικό κόστος στους εργαζόμενους θα έχει σαν αποτέλεσμα μια ελάχιστη βελτίωση για τους καταναλωτές και μια επιδείνωση όχι μόνο στις κοινωνικές συνθήκες αλλά και στις ειδικέ ασφαλείας. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια σε σχέση με τις καταστάσεις των αεροδρομίων και δεν μπορώ με τον τρόπο αυτό να θεωρήσω ότι μια λύση συλλήφδη μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να δούμε καλύτερα την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης περισσότερου ανταγωνισμού και των ζημιών που μπορούν να προκύψουν για τους εργαζομένους αλλά και για τους καταναλωτές. Πολύ ωραία. Εγώ κυρία Πρόεδρε θέλω να δώσω και λίγη μεσογειακή δίαιτα. Λίγο, <laughs> λίγο λάδι, λίγο κρασί γιατί μέχρι στιγμή η συζήτηση είχε κεντροευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θέλω να πω δύο πράγματα με μεγάλη σαφήνεια στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για το, τα μεταφέρει στις, στους προϊσταμένους του. Πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς υπερβολικά συχνά, η Κομισιόν όταν λαμβάνει το χώρο ξεχνά ότι βρισκόμαστε υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας όπου υπάρχει ένα άρθρο 9 που είναι μια ρήτρα που λέει ότι σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής ε, ένωσης θα πρέπει να ε, επιζητηθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητος στην εργασία. Μιλάμε πάντα για το κόστος των, ε, της εργασίας, αλλά δεν λέμε τίποτα για, την, <clears throat> για τις κοινωνικές συνδίκες εργασίας και την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ διαφοροποιημένες θέσεις για αυτά τα θέματα. Πάντα η Κομισιόν βρίσκεται με στο πλευρό των εργοδοτών και είναι πάντα αντίμαχοι με την άποψη των εργαζομένων. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία έκπληξη για το γεγονός ότι ενώπιον των πολιτών, ενώ θα έπρεπε η Κομισιόν να είναι αυτή που είναι ο υπέρμαχος και ο θεματοφύλακας του ευρωπαϊκού υποδείγματος, είναι αυτή η οποία είναι έτοιμη να καταστρέψει και να ακυρώσει ακόμα και τα κεκτημένα που έχουν επιτευχθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ουσιαστικά Μα φέρνει από την πίσω πόρτα η Κομισιόν ένα υπόδειγμα που δεν είναι πια το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και δεν είναι η κοινωνική οικονομία τη αγορά, αλλά είναι απλώ η οικονομία τη αγορά. Εμεί, λοιπόν είχαμε δεχτεί την οικονομία της αγοράς γιατί είχε κάτι το οποίο είχε και ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Αλλά δεν τη δεχτήκαμε μονάχα ξεροσφύρι οικονομία της αγοράς, θελήσαμε να έχει και τον κοινωνικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους που πιστεύουν στην Ευρώπη, στην Ευρώπη των πολιτών, στην Ευρώπη των εργασομένων. Θέλουμε να έχουμε μία Ευρώπη που είναι κοινωνική Ευρώπη. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο θέμα κόστους, είναι θέμα κοινωνικού διαλόγου, είναι θέμα οικοδόμησης συμφωνιών και συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων για να έχουμε καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτηση. Επομένως, θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι τουλάχιστον θα, έχετε ένα, θα πρέπει να ξέρετε ότι από τους σοσιαλιστές βουλευτές τουλάχιστον θα έχετε πολλά προβλήματα με αυτή την πρόταση. Κύριε Σιγητά, θέλετε να θέσετε ερωτήματα συγκεκριμένα στους καλεσμένους μας. Αν ναι, γρήγορα γιατί δεν έχουν χρόνο να απαντήσουν. Νομίζω ότι η μόνη επιταγή την οποία πρέπει να δεχτώ είναι πάντα η επιταγή του περιορισμένου χρόνου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει αν υπήρχε και ένας άλλος πάροχος υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη ποιότητα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να πούμε ότι στα αεροδρόμια εκεί που λειτουργούν τα πράγματα θα πρέπει να έχουμε και ένα παραπάνω πάροχο για να έχει μεγαλύτερη, μεγαλότερο ανταγωνισμό. Θεωρείτε ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μια καλύτερη κατάσταση, θα διατηρηθεί ή θα βελτιωθεί η ποιότητα. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το θέμα της δυνατότητας απασχόλησης των ε, ατόμων στα αεροδρόμια. Λέει η Κομισιόν ότι φτάνουν δύο μέρες απασχόλησης τη βδομάδα. Αλλά είναι δυνατό να το δεχτούμε αυτό. Κάποιος ο οποίος εξυπηρετεί ένα αεροπλάνο και έχει μία κατάρτιση ειδική για τα θέματα αυτά. Αν βιδώσει λάθος μια βίδα, μπορεί να πέσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, κάπου πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη και θα ήθελα να ξέρω να ποιες είναι οι απόψεις των τριών σας για το θέμα αυτό. Και μετά το θέμα το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος Χέντελ για τα εισιτήρια, ότι αναφερόμαστε μονάχα για 1,6 ευρώ που θα κερδίσουμε σε ένα εισιτήριο 200 ευρώ και για να το πετύχουμε αυτό καταστρέφουμε και εξολοθρεύουμε ένα ολόκληρο εργασιακό τομέα. Είπε σαφώς και ο κύριος ε, Σέρκας ότι δεν είναι θέμα βορρά ή νότου, είναι θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Και το τελευταίο στοιχείο αναφέρθηκε, είναι το θέμα του πώς είναι οι εργαζόμενοι. Αναφέρθηκε από τον κύριο Κιόπχεν δεν είναι 60.000 αλλά ότι είναι 300.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε βέβαια περιορισμένες αρμοδιότητες για το άρθρο 6 αλλά εμείς ως μέλη της Επιτροπής ε, Απασχόλησης μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Το, η δική μου έκθεση εστιάζεται μονάχα στους δικούς μας τομείς για θέματα που είναι προαιρετικά ή υποχρεωτικά, αλλά μπορούμε να υποβάλουμε και τροπολογίες και για τα θέματα που δεν είναι στενά της Επιτροπής μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Σύμφωνα απολύτως. Στον φάκελο αυτόν αν δούμε και το χάρτη που μας ε, μοιράσετε, η Γερμανία και η Ελλάδα ε, είναι ενωμένε στο ίδιο μέτωπο. Δίνω τον λόγο στους προσκεκλημένους μας. Σας προτείνω να σας ακούσουμε με την ίδια σειρά. Δυστυχώς ε, έχετε πέντε λεπτά το πολύ ο καθένας για να μπορέσετε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Εξαιρετικά εύστοχες, με βάση την εμπειρία μου θα προσπαθήσω να δώσω τις πληρέστερες δυνατές απαντήσεις. Πέντε σημεία κατέγραψα. Το κόστος καταρχήν. και είναι οι επιπτώσεις του κόστους των υπηρεσιών στην τιμή του ειστηρίου. Εμείς ως αεροπορική εταιρεία ξέρουμε ότι οι υπηρεσίες επίγειες εξυπηρέτησης είναι στοιχείο κλειδί στην αντιγωνιστικότητά μας, διότι υπάρχει αμέσως αποτέλεσμα το αποτέλεσμα. Το 15% που σας έδωσα δεν είναι μόνο οι αποσκευές και η καθοδήγηση των αεροσκαφών, αλλά είναι και άλλες ε, υπηρεσίες, ε, τα σαλόνια αναμονή των επιβατών, άλλες υπηρεσίες επιβατών κλπ. Γι' αυτό είπα 15% και 15% είναι πολύ. Στο παρελθόν ε, ξέρουμε ότι μειώθηκαν οι δαπάνες αυτές, όμως ε, σιγά σιγά τελευταία βλέπουμε και μεγάλες διαφορές στην εξυπηρέτηση ενός αεροσκάφους. Ε, αλλού είναι 2.000, αλλού είναι 400 μόνο ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι με σταδιακή επελευθέρωση, λελογισμένη, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλο φαλή για τις αεροπορικές εταιρείε. Είναι υπηρεσίες, επίσης, απαντώ και στο ερώτημα αυτό, κλειδί. Ναι, είναι για μας, διότι επηρεάζουν τα αποτελέσματα, επηρεάζουν ακόμη και την ακρίβεια στην παράδοση των αποσκευών, την ακρίβεια των δρομολογίων και ούτω καθεξής. Από όλα αυτά και εμείς κρινόμαστε. Εξαρτώμεθα από τις υπηρεσίες. Αν κάτι δεν πάει καλά εκεί, οποιοδήποτε λεπτό καθυστέρησης για μας κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ. Το λεπτό. Οπότε λοιπόν, ναι, οι υπηρεσίες αυτές είναι κρίσιμε για τι αεροπορικέ εταιρείε και πιστεύουμε ότι μειώνοντα το κόστος των πηγών υπηρεσιών εμέσως ή εμέσως, χωρί να απομειωθεί η ποιότητα, μπορούμε να μειώσουμε το εισιτήριο κατά παραπάνω από ένα ευρώ. Ακούστε και κάτι άλλο από συναδέλφους και βουλευτές. 70-80% του κόστου των υπηρεσιών είναι κόστο προσωπικού. Αυτό είναι σωστό. Αυτό γνωρίζουμε και εμεί από την πείρα μα. Όμω, μείωση του κόστου δεν σημαίνει μείωση των μισθών αναγκαστικά. Καλές εταιρείε στον τομέα βελτιώνουν την απόδοση των εργαζομένων, τους συνδυάζουν σε διαφορετικές λειτουργίες και καθήκοντα, προσαρμόζονται σε απαιτήσει των πελατών. Προφανώς ο μισθός είναι παράμετρος, αλλά δεν είναι η μόνη παράμετρος που επηρεάζει το τελικό κόστος. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να συνδυάσουμε την εμπειρία από διαφορετικά αεροδρόμια, να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές, να ανέβει η απόδοση. Αυτοί είναι οι τρόποι και όχι αναγκαστικά να μειωθούν οι μισθοί. Το θέμα είναι λοιπόν να γίνουμε πιο επαγγελματίες στον τομέα μας. Τρίτον, αν δείτε την κατάσταση σήμερα στα αεροδρομία της Ευρώπης, ε, δύο είναι μεγάλοι και αυτό δεν είναι καλό για τον ανταγωνισμό προφανώς. Παρ' όλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα αεροδρόμια, είναι δύσκολο για μεγάλες αεροπορικές εταιρείε να αφήσουν τον, τη μία εταιρεία και να πάνε στην άλλη λόγω του κόστου της μετάβασης. Και υπάρχει και ένας κίνδυνος. Υπάρχει σχεδόν υποχρέωση, είναι, είναι ανάγκη θα έλεγα, από δύο εταιρείε να πάμε σε τρει στα μεγάλα αεροδρόμια. Οι Βρυξέλλες είναι ένα παράδειγμα και το ίδιο υποστηρίζει και η Star Alliance. Σε μεγάλα αεροδρόμια λοιπόν για τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείε, δύο εταιρείε πηγή εξυπηρετή σημαίνει ουσιαστικά μονοπόλιο. Εκεί που υπάρχουν δύο εταιρείε μόνο βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν εταιρείε οι οποίες κατά τα άλλα τηρούν την εργατική νομοθεσία, σέβονται τους υπαλλήλους τους αλλά δυστυχώ αναγκάζονται πολλέ φορέ να αποχωρήσουν, να σταματήσουν την παροχή γιατί δεν υπάρχει αρκετή δουλειά. Από τη δική μα εμπειρία και από συζητήσει που έχουμε με άλλου ε, παρόχου και άλλε αεροπορικέ εταιρείε, δεν είμαστε υπέρ του ανεφόρων όρων ανοίγματο οποιοδήποτε αεροδρομίου. Όχι. Το άνοιγμα πρέπει να γίνει σταδιακά, λελογισμένα, προσεκτικά, από δύο σε τρει καταρχήν εταιρείε, για να μπορέσει να βελτιωθεί καταρχήν η ποιότητα. Αν αυτό γίνει προσεκτικά, παραλαμβάνω, θα βελτιωθεί και η ποιότητα. Και κύριε Πρόεδρε, ε, δύο παραδείγματα αεροδρομίων. Όχι, σα ευχαριστώ, ε, λέει πρόεδρο. Πρόεδρος. Κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι μέλος διοικητικών συμβουλίων δύο επιχειρήσεων. Μεσαίων επιχειρήσεων που είναι του μεγέθους της ε, Brussels Airlines. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία και είναι περίπου τα ίδια. 850 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συνολικό κόστος που περιλαμβάνει λειτουργικό κόστος, αεροσκάφη, ασφάλειες κτλ. Από αυτά τα 85 εκατομμύρια, 9% περίπου, 40 εκατομμύρια είναι το κόστος ε, εξυπηρέτησης εδάφους. Αλλά αυτό είναι το κόστος για υπηρεσίες οι οποίες όχι μόνο κόστος το οποίο είναι η υπορρύθμιση στη Γερμανία, αλλά και στοιχεία κόστους τα οποία βρίσκονται εκτός του τομέα ρύθμισης. Αν λάβει κανείς υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, βλέπετε ότι είναι στην, ε, το κόστος της εργασίας της τάξης του 60 με 80%. Και βλέπουμε, πιστεύω ότι άμα τα δει όλα αυτά, το κόστος της εργασίας δεν ε, ξεπερνάει το 0,3% του συνολικού κόστους και μπορεί κανείς να δει ότι σε μια πτήση η οποία κοστίζει 400 ή 200 ε, ευρώ ποιο είναι το τμήμα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την, ε, με την εργασία. Για μια μεγάλη εταιρεία Μπορεί το κόστος αυτό να είναι κάποια εκατομμύρια, αλλά προ, ε, προκαθορίζει και περαιτέρω την ε, περαιτέρω κέρδη και ίσως και την αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά δεν αλλάζει το πραγματικό κόστος των ε, πτήσεων ή του, των ναύλων. Και πιστεύω ότι στις Βρυξέλλες υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι πολύ καλά ε, οργανωμένες. Η Lufthansa έχει παρουσιάσει τα στοιχεία της πολλές φορές στο παρελθόν και έχει δείξει ότι το κόστος της εξυπηρέτησης εδάφους δεν ξεπερνάει το 4,4 του συνολικού κόστους για, τις δεύτε, για το δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Υπάρχει μια μελέτη η οποία ασχολείται με το κόστος της εξυπηρέτησης εδάφους για τις αεροπορικές εταιρείε, ώστε να μην βασιζόμαστε μονάχα σε ε, υποκειμενικές απόψεις που διατυπώνουμε εμείς. Τι θα γίνει αν η Κομισιόν περάσει την πρότασή της ή ακόμα και να αποχωρήσει και περισσότερο από αυτά. Τότε το αποτέλεσμα θα είναι ότι σε χώρες όπως η Αγγλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία να επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες. Και αυτό θα αφορά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες όπου υπάρχουν ακόμα περιορισμοί θα επιταχυνθεί η επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών και της κατάρτισης ο κύριος μίλησε για την ε, εκπαίδευση που υπάρχει σε πολλές θετικές εταιρείες εξυπηρέτησης. Ακόμα και οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν την κατάρτιση των εργαζομένων. Όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, έχουν επίπτωση πάνω στην ε, ασφάλεια. Αν δούμε λοιπόν το επίπεδο αποδοχών των ε, επιχειρήσεων αυτών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί κανείς να φανταστεί πού θα φτάσουν, πόσο χαμηλά θα κατέβουν αυτές οι αποδοχές όταν δεν υπάρχουν κοινωνικές ε, ρήτρε και θα υπάρξει μεγαλύτερη φιλεδροποίηση Τελικά ο φορολογούμενο όλο και περισσότερο πρέπει να πληρώνει το κόστο τη απώλεια θέσεων εργασία και τα επιδόματα ανεργία. Δεν κερδίζει τίποτα με τον τρόπο αυτό. Κανεί μα δεν θέλει κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι ανεξάρτητα από το αν έρχεται κανείς από την Αγγλία, από την Ελλάδα, την Πορτογαλία ή την Πολωνία, όλοι έχουν κοινό συμφέρον αυτός ο ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας των εναρίων μεταφορών να λειτουργεί σωστά και θα πρέπει οι εργαζόμενοι εκεί να έχουν ε, την εξασφάλιση ότι η εργασία τους καλύπτεται από αυτά που λέει η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν θα πέσουν θύμα κάποιων ε, επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μεταβλητή επί τη βάση του κέρδους αποζημίωση. Μάλιστα, ο τελευταίος μας προσκεκλημένος. Ο κύριος Κόψεν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολύ καλές σας ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο αεροδρόμιο της Βιέννης. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο αλλά μπορώ να πω ότι να μιλήσω για τα αεροδρόμια που έχουν πραγματικές υπηρεσίες εδάφους, ε, θα δείτε ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια σε ε, ε, το ερώτημα που πρέπει να τεθεί όσον αφορά την περαιτέρω απελευθέρωση είναι πώς μπορεί να υπάρχει ε, μεγαλύτερο κέρδος για τα αεροδρόμια αυτά. Ε, γιατί η απελευθέρωση θα έχει κάποιο αντίκτυπο και ε, στο κέρδος για τα αεροδρόμια. Τώρα για το ερώτημα τώρα της ε, άθεσης του προσωπικού πρέπει να το δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα γιατί ορισμένοι μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι μιλάμε για ε, γερμανικά ζητήματα ή τέλο πάντων για θέματα που αφορούν ε, συγκεκριμένες χώρες. Όχι, μιλάμε για έναν κανονισμό που θα ισχύει για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 27 και αυτά τα οποία αναφέρω εγώ αφορούν όλα τα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το θέμα συγκεκριμένα που αφορά το προσωπικό, ε, ένα δείγμα είναι η Ισπανία, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία ε, για τη μετάθεση και Άλλες χώρες έχουν πολύ πιο περιορισμένη ε, πρόσβαση στην αγορά. Το να είναι λοιπόν δεσμευτικό αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τις ίδιες τις χώρες και δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο ή τέλος πάντων μετά από κάποιο χρόνο ε, που θα έχει περάσει ε, από τη μετάθεση ε, θα μπορούσε μετά πάλι ο εργοδότης να τον απολύσει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι επαρκές επιχείρημα κατά της συγκεκριμένη διάταξης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ένας μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας για το προσωπικό αυτό. Ε, αν λοιπόν απελευθερωθούν οι αγορές έτσι όπως το προτείνουμε, 7 χρόνια είναι τουλάχιστον ο χρονικός αυτός ορίζοντας. Διαφορετικά μπορεί κανείς να χάσει τη δουλειά του. Είναι λοιπόν σημαντικό, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια της απασχόλησης για τους εργαζόμενους αυτούς. Χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται ποιότητα για τις υπηρεσίες. Δεν θέλουμε να χάσουμε την τεχνογνωσία των ανθρώπων αυτών. Δεν μιλάμε για μια πλήρω απελευθερωμένη αγορά, γιατί τότε είναι αλλιώ τα πράγματα. Εγώ μιλάω για το άρθρο 12 που αφορά συγκεκριμένα ε, κάποιους ε, κάποιες αγορές που έχουν απελευθερωθεί αλλά με κάποιους περιορισμούς. Τώρα, η εξυπηρέτηση εδάφους με ίδια μέσα. Η αυτοεξυπηρέτηση. Ε, είδαμε τη δυνατότητα απεργολαβία από πλευρά αεροπορικών εταιριών, κάτι το οποίο έχει τεράστια, ε, τεράστιο αντίκτυπο από κοινωνική απόψεω. Δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιε. Ή οι κάνουν αυτή τη δουλειά ή ε, προβαίνουν σε υπερβολαβία. Αν αλλάξουμε τον ορισμό και επιτρέψουμε την υπεργολαβία, τότε θα μπορούν να βρουν ένα τρίτο ε, ε, φορέα, οι αεροπορικές εταιρείες, που μπορεί να μην είναι ένας από τους ε, δύο, ε, τρεις που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη περιορισμένη αγορά. Οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα υπάρξει μεγαλύτερη πίεση και, για, και στις τιμές και στις κοινωνικές συνθήκες. Δεν μιλάμε μόνο για μία χώρα, για τέσσερις χώρες το θέμα του ανοίγματο τη αγορά, το θέμα της αυτοεξυπηρέτησης είναι, και του ορισμού του ε, αφορούν όλα τα κρατημέλη όπως και οι ε, κοινωνικές συνέπειες ε, των διατάξεων αυτών. Το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μαν ε, κατά πόσο ένας επιπλέον φορέας ε, ε, θα έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα εξαρτάται από το αεροδρόμιο. Υπάρχουν αεροδρόμια που έχουν τρεις-τέσσερις εταιρείε και έχουν πολύ καλό, καλή ποιότητα και δεν δημιουργεί πρόβλημα κάτι τέτοιο. Όμως μερικές φορές δεν υπάρχουν οι συνθήκες της αγοράς για να υπάρξει τρίτος φορέας ας πούμε αν ε, μια αεροπορική εταιρεία έχει το 70% του όγκου της κυκλοφορίας ε, και ε, υπάρχει μια τρίτη εταιρεία που ασχολείται με το υπόλοιπο 30% τότε τι γίνεται υπάρχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά διατηρείται η ποιότητα σε ορισμένα αεροδρόμια ε, λοιπόν υπάρχει ε, περιθώριο περιτέρου ανοίγματο και είναι καλή ιδέα, σε άλλα αεροδρόμια δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώ είπα ότι είναι καλύτερα να δούμε τι τοπικέ συνθήκε, ε, να υπάρχει δηλαδή μια διακριτική ευχέρεια για τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει σε κάθε κράτο μέλο πόσο θα ανοίγει η αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επίση να λάβει το λόγο και θα ήθελα να του ζητήσω να είναι σύντομη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ε, δευτερολογήσω. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, εμείς καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο πολιτικό και πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το ζήτημα. Έχουμε λάβει υπόψη ε, όλα αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα τα σημειώνουμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρότασή μα πρέπει να είναι εξισορροπημένη, πρέπει να λαμβάνει πλήρω υπόψη την ε, κοινωνική διάσταση και συμφωνώ απολύτω με αυτά που είπατε κύριε Σέρκας σε σχέση με αυτό. Γι' αυτό η πρότασή μα είναι εξισορροπημένη και γι' αυτό συμπεριλαμβάνει αυτές τις βασικές διατάξεις ε, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορούν να το κάνουν λόγω των ε, κρεμών δικαστικών υποθέσεων να μπορέσουν να ανοίξουν κάπως την αγορά τους. Χωρίς αυτόν τον κανονισμό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την απελευθέρωση όμως ο κανονισμός αυτός. Η απελευθέρωση που προτείνουμε είναι πολύ περιορισμένη. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε η Brussels Airline για, την σταδιακή, για τη σταδιακή ε, προσέγγιση που αφορά πολύ συγκεκριμένους τομείς ε, που δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός και λέμε να μπορούμε να περάσουμε από δύο σε τρει παρόχους μόνο στα μεγαλύτερα αεροδρόμια. Κάτι ακόμη κυρία Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν πολλά για την εκπαίδευση εκπαίδευση, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι μεγάλη σημασία. Είναι γεγονός ότι λιγάκι έχει παραγνωριστεί αυτό το θέμα στον κλάδο αυτών. Ε, πιστεύουμε ότι η ανάγκη υποχρεωτική εκπαίδευση υπάρχει και γι' αυτό έχει, αυτό έχει άμεση σχέση με τι προδιαγραφέ ποιότητα. Πολύ καλά τα σχόλια που ακούστηκαν από αυτού. Κυρία Στάινχαρτ, αναφερθήκατε, Στάινρουξ, ε, αναφερθήκατε κυρίω ε, στο θέμα τη ασφάλεια. Βεβαίω πρέπει να καλύπτεται από τι προδιαγραφέ ποιότητα. Και αυτό εννοώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε λοιπόν προς το παρόν για το πρωί. Και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν εξετάσουμε το σχέδιο γρομοδότησης του κυρίου Τόμας Μαν στις 20 Ιουνίου. Στις 3 ώρες συνεχίζουμε.